της υποεπιτροπής μας φέτος. Παρακαλώ να κάνετε ησυχία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Είναι μια χρονιά η οποία ε, θα έχει τεράστια σημασία για την υποεπιτροπή μας από τη στιγμή που το θέμα της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό ως εξέλιξη. Το Κοινοβούλιο βεβαίως δεν είχε προσυπογράψει πλήρως ε, την ε, άγουσα, όμως ε, πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε, θέλουμε να συμβάλλουμε, γι' αυτό και θα οργανώσουμε διάφορες ακροάσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ώστε να ακούσουμε τη μαρτυρία εγνωσμένων προσωπικότητων στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, έτσι ώστε να μπορέσουμε καλύτερα να διαμορφώσουμε τις θέσεις μας, τις πεπιθήσεις μας για να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας πόσο μάλλον σήμερα με την κρίση του Μαλή ε, που φαίνεται πόσο αδύρυτη ανάγκη είναι να έχουμε μια τέτοια πολιτική. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται διαδικτυακά και θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να ε, εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Ζουλιαν ε, Αχμαν Ζουλιά, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας μέχρι ε, τις 31 του 12 του 12 και ο οποίος συνταξιδοτήθηκε, σίγουρα μας παρακολουθεί διαδικτυακά. Η κυρία Βόλτερ Ντρόπ τον αντικαθιστά, την ευχαριστώ θερμά προσωρινά τον αντικαθιστά και έτσι έχουμε εκπρόσωπο από τη Γραμματεία για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Έχουμε τρεις προσκεκλημένους σήμερα. Ο καθένας θα μιλήσει για, διαφορετικό θέμα. Ωστόσο, θα ακούσουμε πολύ σημαντικά πράγματα από πολύ σημαίνουσες προσωπικότητες με ε, αδιαφυσβήτητη εμπειρία. Ο πρώτος που μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας είναι ο στρατηγός κ. Νόμαντ, ο οποίος είναι πασίγνωστος από τους ειδικού, τους εμπειρογνώμονες και όχι μόνο. Δεν θα αναφέρω το σύνολο της σταδιοδρομίας σας ε, στις ε, γερμανικές ε, στρατιωτικές ένοπλες δυνάμεις. Ήσασταν αρχηγός του Γερμανικού Στρατιωτικού Επιτολίου, πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ από το 1996 μέχρι και το 1999. οπότε και είχαν γίνει πολύ σημαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις από το ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, στα Βαλκάνια, γεγονότα τα οποία θυμόμαστε βεβαίως όλοι. Ε, αξιοποιώ αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω και τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Πέτερινγκ, ο οποίος έχει προεδρεύσει σε αυτή την υποεπιτροπή, χάρη στον οποίο άλλωστε Έχουμε την τιμή να υποδεχόμαστε τον στρατηγό κύριο Νόμαντ μαζί μας σήμερα. Δεν θα χρονοτριβήσω παρακαλώ, στρατηγέ έχετε το λόγο. Euh, ευχαριστώ Πρόεδρε, Σα ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είναι πραγματικά τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ και συζητώ μαζί σα τις μελλοντικέ επιλογές για βελτιωμένε δυνατότητες άμυνα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, και του ΝΑΤΟ. Μου είπαν ότι μπορώ να μιλήσω γερμανικά και γι' αυτό θα ε, μιλήσω στην μητρική μου. Χαίρομαι ιδιαίτερος που ως πρώην και πρώτος ε, ε, γραμματέας ε, του Γαλλογερμανικού Συμβουλίου για την Ασφάλεια και την Άμυνα. Σήμερα, μία μέρα μετά από την 50η επέτειο της Συνθήκης των Ηλυσίων, έχουμε εδώ τη δυνατότητα να συζητήσουμε τις ιδέες ε, της δημιουργίας ε, μιας ευρωπαϊκής ε, δύναμης η οποία θα εξυπηρετήσει την πρόθεση της ευρωπαϊκής άμυνας. Το σημείο αφετηρίας της πρόσκλησής μου εδώ ήταν δύο ερωτήσεις σε συναδέλφους σας, τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Πέτερινγκ. Ε, τον ρώτησα εάν ε, θα μπορούσε να φανταστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τη δυνατότητα, εφόσον η Κομισιόν έχει περιορισμένες δυνατότητες για την περιοριστική άμυνα αν θα μπορούσε με βάση κάποιες προϋποθέσεις να ζητήσει από την Κομισιόν να επεξεργαστεί τελικά την πολιτική ασφάλειας για το 2013 στην αναθεωρημένη μορφή του 2008 και μετά σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν για αλλαγές και τη χρήση της στρατηγικής. Επίσης τον ρώτησα αν θα ήταν δυνατό να φανταστεί το Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Κομισιόν να προωθήσει την ιδέα όλα τα κράτη ε, που ε, έχουν τη συμβολή τους ε, στην κοινή πολιτική να δεσμευτούν να αυτά τα, τα, αυτές τις μονάδες που έχουν να τις χρησιμοποιήσουν από κοινού επειδή είχα στο μυαλό μου ότι κάθε φορά υπάρχει επιφύλαξη κοινοβουλευτική εξέταση στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, η οποία πάντοτε καθυστερεί τη διαδικασία, ε, ήθελα να δω αν ε, κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να αποφευχθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, συχνά λοιπόν ε, στο ΝΑΤΟ, όπως έχω δει ε, στο παρελθόν, κάτι τέτοια πράγματα είναι πιο εύκολα. Ο κύριος Πέτερινγκ θεώρησε πολύ ενδιαφέρουσα την ερώτησή μου και σας ε, πρότεινε κύριε Πρόεδρε να με καλέσετε εδώ και να με. Το σημείο αφετηρίας των ερωτήσεων μου είχε να κάνει κυρίως με την κακή κατάσταση των ευρωπαϊκών δυνάμεων άμυνας. Τα ευρωπαϊκά κράτη ε, δίνουν γύρω στα 200 δις ευρώ το χρόνο για την άμυνα και έχουν περίπου 1,7 εκατομμύρια στρατιώτες που είναι περίπου το 40% των ε, δαπανών των Ηνωμένων Πολιτειών και σχεδόν 200.000 άντρες περισσότεροι από αυτούς που διαθέτουν ε, οι Αμερικανοί. Όμως, όταν, υπάρχει, όταν υπάρχουν αποστολές σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Ευρωπαίοι έχουν μόνο το 10% της δυνατότητας εμπλοκής των Αμερικάνων. Από τη στιγμή βέβαια που συμφωνήσουν 27 κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια τους. Εφόσον συνεχίζει αυτή η κατάσταση, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άποψη, δική μου άποψη, ε, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κρίσεις από μόνη της ε, και σε μια εποχή πολλών κρίσεων και σειράξεων είναι πιο εξαρτημένοι από τη ΣΥΠΑ από ότι ήταν κατά τον ψυχρό πόλεμο. Οι Αμερικανοί στρέφονται προς την Ασία και προς το συμφέρον των Ευρωπαίων και το κάνουν επειδή πρέπει, αλλά θα μπορούσαν ως μεγάλη ναυτική δύναμη αν η άλλοι ε, όχθη αυτή της Ευρώπης και η γύρω περιοχή ε, ήταν οι ήσυχοι μόνο τότε θα μπορούσαν να το κάνουν. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και θα φανεί και στο μέλλον σύντομα από τη Λιβύη και από το Μαλί όπου μόνο η Γαλλία με τη βοήθεια των Δυτικοαφρικανών δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Έτσι λοιπόν η, η Ευρώπη δίνει χρήματα σε εθνικά προγράμματα και εξοπλίζεται για τον πόλεμο του χθες, χρησιμοποιεί πολύ λίγο την παγκόσμια αγορά και συχνά θεωρεί ότι ενισχύει την βιομηχανία εξοπλισμών όταν στην ουσία απλώς επανεφεύρει τροχούς και οι Ηνωμένε Πολιτείε ήδη έχουν περάσει στην παραγωγή των επόμενων ε, μοντέλων. Τι πρέπει να κάνουμε. Το να συνεχίζουμε έτσι ή το να χρησιμοποιούμε έτσι κοσμητικές ε, εκφράσεις όπως το pooling και sharing κοινή χρήση και των δυνάμεων ε, δεν πρέπει να ε, είναι πλέον ε, μέσα στις προτάσεις, όπως είπε ήδη η Βαρόνια Άστον στο Σεπτέμβρη στο Συμβούλιο. Πρέπει τα ευρωπαϊκά κράτη να συνεργαστούν μεταξύ τους ακόμα πιο στενά, να αφήσουν στην άκρη κομμάτι της εθνικής τους κυριαρχίας και για κάποιες αποστολές ε, που ε, είναι από οικονομική άποψη λογικό να τις κάνουν από κοινού ε, και να χρησιμοποιούν μονάδες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα χρηματοδοτούνται και από αυτήν. Σκέφτομαι τις κατηγορίες Enabler και Force Multiplier. Αυτό θα σήμαινε ότι τα κράτη δεν θα αντρούν εθνικά σε αυτό το επίπεδο και γι' αυτό θα πρέπει να δεσμευτούν να έχουν μονίμως ε, τέτοιες μονάδες όταν, ε, και να τις χρησιμοποιούν όταν απαιτείται. Για να διατηρήσουν τα δικαιώματα των Εθνικών Κοινοβουλίων μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα, ε, να δημιουργηθεί το Component Forces της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα παίρνει έγκριση από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έτσι θα μπορεί να δράσει η Ευρώπη όπως και δρούν και οι ΕΕ. Και θα ήταν καλό αυτά τα components να έχουν την εξής δομή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει κομμάτια τα οποία θα έχουν τον ίδιο εξοπλισμό και την ίδια εκπαίδευση όπως και τα αμερικάνικα components τα οποία σε επίπεδο ΝΑΤΟ ε, χωρίς καμία καθυστέρηση μπορούν να δημιουργήσουν μια γενικότερη δύναμη ε, που θα περιλαμβάνει όλα τα components ε, σύμφωνα με τα πρότυπα των AWACS και του, της αποαέρωσης επιτήρησης του πεδίου. Έτσι, Έχουμε με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές ε, ενοπλές δυνάμεις ε, ε, θα είναι ο πρόδρομος ενός ευρωπαϊκού στρατού μια τέτοιας υποτοπικής ιδέας, αλλά θα έχουμε από κάτω προς τα πάνω μια μεγάλη δυνατότητα να έχουμε ευρωπαϊκές συνολικές δυνάμεις. Τι εννοώ η Ευρώπη θα μπορούσε να έχει την EU Mail Component Force, μία από κοινού χρηματοδοτούμενη και λειτουργούμενη μονάδα που θα συμπληρώνει την AGS Component Force του ΝΑΤΟ. Δηλαδή ένα mail το οποίο θα μπορεί να επανδρώνεται ε, και να πετά όπως ένα Firebird και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο υπάρχουν ε, ε, διάδοχοι των AWACS ε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να έχουμε κοινή ανάπτυξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Οργανισμός για τη Διαχείριση των Μαχών θα ήταν επίσης σε επίπεδο αντιπριλαβλικής άμυνας ένα παράδειγμα δυνατό. Φυσικά ε, πρέπει πάντοτε να έχουμε ε, εργασία από κοινού, αλλά και σε επίπεδο θαλάσσιων μεταφορών ή σε μια αερομεταφερόμενη τέτοια μονάδα ευρωπαϊκού επίπεδου, που θα είχε και την συνδρομή δυνάμεων της NL Rotterdam, του επίπεδου του NL Rotterdam, ε, θα μπορούσαμε να έχουμε και διάφορα μεταγωγικά τα οποία θα ήταν ιδανικά εργαλεία. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες τότε θα μπορούσαμε να έχουμε, για παράδειγμα, ένα ελικόπτερο βαρέων μεταφορών ως ε, διάδοχο του CH-47 και του CH-53, το οποίο ε, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τις δυνάμεις του Ρότερνταμ ε, και να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σε κρίσεις ε, και σε ανθρωπιστικές καταστροφές που λόγω της ε, κλιματικής αλλαγής όλο και περισσότερο θα βλέπουμε. Ένα... Έτσι λοιπόν ένα από τα πράγματα που ισχύει είναι ότι το 80% των περιοχών που χρειάζονται την ε, συνδρομή μας είναι πολύ μακριά από τις ακτές. Ένα παράδειγμα επίσης ενός force multiplier είναι μια δυνατότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αεροπορικές επιθέσεις. Δεν σκέφτομαι τόσο το FPA, αλλά το EU UCAV Component Force, το οποίο θα είχε το πλεονέκτημα ε, να, για τις... Ε, όταν χρησιμοποιείται να μην χρειάζεται ούτε staging ούτε overflight. Τέτοια δικαιώματα δηλαδή υπερπτήσεως ε, και ε, ανάπτυξης. Σε κρίσεις χρειάζεται να δρούμε γρήγορα και όταν υπάρχουν ε, συνεχώς διαπραγματεύσεις τότε δίνουμε ένα εργαλείο στα χέρια των εχθρών. Μέσα λοιπόν από την ενίσχυση της δυνατότητας δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μην υπάρχουν σειράξεις ε, στις οποίες ε, θα πρέπει να δρούμε από μόνοι μας. Έχουμε το πλεονέκτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση άτο του ΝΑΤΟ ότι έχουμε και πολιτικά μέσα ένα από τα πρώτα βήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την κατεύθυνση ήταν ε, οι ευρωπαϊκές αστυνομικές δυνάμεις. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχουμε γρήγορα χρησιμοποιούμενες δυνάμεις για την ε, αντιμετώπιση καταστροφών, ειδικότερα σε Τομεί, όπω ο βιολογικό, χημικό, πυρηνικό πόλεμο κτλ. Ω Ευρωπαίοι λοιπόν αναρωτιέμαι γιατί μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι δικές του ένοπλε δυνάμει έχουν εδώ και καιρό ε, τη δυνατότητα να έχουν στολές που τους προστατεύουν σε τέτοια περίπτωση ενώ εμείς δεν έχουμε. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα στη Γερμανία να φτιάξουμε τέτοιες στολές και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε ως προστατευτικές στολές σε περίπτωση βιολογικού, χημικού κτλ. πολέμου. Και θα ήταν καλό το Κοινοβούλιο να ζητήσει τελικά οι Ευρωπαίοι ε, στρατιώτες να έχουν τη δυνατότητα μιας τέτοιας στολής. Δεν μπορώ τώρα να σας δώσω άλλα παραδείγματα, αλλά θα έλεγα ότι με βάση και το δικό σας ενδιαφέρον θα ήταν καλό να υπάρχει μια νέα αναδιατύπωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας με συγκεκριμένες ε, ε, διατάξεις που θα δίνουν το βάρος ε, στην ευρωπαϊκή δράση και θα προωθούν τα συμφέροντα της Ευρώπης, όπως ας πούμε ζήτησε και η Άστον, ε, έτσι ώστε να έχουμε διαλειτουργικότητα μετα, ε, μεταξύ ΝΑΤΟ και των δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ε, την κατάσταση έτσι ώστε να μπορούμε να δρούμε στο πεδίο του μέλλοντος. Και με βάση την έρευνα και την ανάπτυξη και τον συντονισμό στο πεδίο να μπορούμε να ε, δρούμε, για παράδειγμα, σε τομείς όπως η νανοτεχνολογία, η ρομποτική και η βιονική. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μου δώσατε και για το χρόνο σας. Ε, ελπίζω να σας έδωσα κάποια πράγματα για να σκεφτείτε και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Είμαι ανοιχτό σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η απόψη σας ε, είναι βεβαίως πάρα πολύ ενδιαφέρουσας, ενδιαφέρουσες και είναι και καρπός ε, της πολύ πλούσιας εμπειρίας σας. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμες για εμάς. Άλλωστε, πολλές από τις απόψεις σας ακολουθούν ε, τις κατευθύνσεις που θέλει να προωθήσει η υποεπιτροπή μας. Ε, βέβαια, είναι δύσκολο να εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη, αυτό πάντοτε ισχύει. Εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση η οποία ίσως έχει περισσότερο σχέση με την ε, γερμανική άποψη για την άμυνα και ίσως θεωρηθεί λίγο προκλητική ερώτησή μου, το κάνω όμως για, να, ε, για το καλό της συζήτησης. Λέγεται συχνά βεβαίως ότι η Γαλλία και η Γερμανία είναι η κινητήρη μοχλή για, την, ε, για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και για την οικοδόμηση μιας πολιτικής άμυνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέγεται ότι δεν μιλούν την, την ίδια γλώσσα στα αμυντικά θέματα. Όταν μιλούν για την άμυνα οι Γάλλοι εννοούν τις επιχειρήσεις ε, και ε, τη θεσμική κατοχήρωση και οι Γερμανοί, οι Γερμανοί μιλούν για τη βιομηχανία, το βιομηχανικό σκέλος, για το οικονομικό σκέλος αν θέλετε της πολιτικής άμυνας. Ε, εσείς συμμερίζεστε αυτή τη γενίκευση, αυτή την απλούστευση. Ε, ποια είναι η γνώμη σας, ποια είναι η γερμανική άποψη, ο γερμανικός τρόπος, αν θέλετε, με τον οποίο ερμενεύεται στη Γερμανία η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Η δυσκολία στην οποία προσκρούμε είναι η εξής. Πάρα πολύ εξημών κάνουμε την εξής διαπίστωση. Εάν δεν σημειώσουμε πρόοδο, και βέβαια πρέπει με μεγάλη προσοχή ε, να τα φροντίζουμε όλα αυτά, αλλά εν πάση πτώση αν δεν μοιράσουμε τα βάρη δεν θα τα καταφέρουμε. Και κάθε φορά που ε, τίθεται το θέμα του μοιράσματος των ε, βαρών, τότε τίθεται και το σκέλος το βιομηχανικό, του κλάδου, της οικονομίας και άρα ε, εκεί προκύπτουν και όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την εργασία, με την απασχόληση, με πάρα πολλά θέματα και άρα εκεί προκύπτουν και ε, οι εκάστοτε εθνικοί εγωισμοί αν θέλετε. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο χωρίς να τρομάξουμε τις χώρες που θεωρούν ότι το κόστος το κοινωνικό ή το εργασιακό, το οικονομικό θα ήταν δυσβάσταχτο. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που θα ήθελα να σας θέσω, αλλά πάρα πολλοί συνάδελφοι θέλουν το λόγο επίσης. Ε, πρώτον ο κύριος Γκάλερ, συντονιστής από το ΕΛΚ για τα θέματα τα αμυντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, στρατηγέ Νόμεν. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή σας. Ε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και για τον τρόπο που μας παρουσιάσετε τα πράγματα. Πραγματικά έχουμε πάντοτε ανοιχτές πόρτες στις θέσεις σας και νομίζω ότι με χαρά ακούσαμε τα όσα είπατε. Θέσατε ε, τα προβλήματα ξεκάθαρα και Ουσιαστικά είπατε ότι αν θέλαμε θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα από κοινού. Το θέμα ε, είναι αν γίνει κάτι οξύ, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που ε, ήδη έχει δημιουργήσει τόσες δομές και παρόλο που έχει δυνατότητες ήδη έτοιμες, γιατί τελικά όταν τα πράγματα γίνονται σοβαρά πηγαίνουμε σε άλλες δομές και ε, προστρέχουμε σε αυτές αντί για τις ευρωπαϊκές. Το μαλλι είναι ένα τρέχον παράδειγμα που πραγματικά απορώ γιατί δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις ε, οι οποίες θα μπορούσαν να προχωρήσουν από τα κράτη-μέλη από κοινού και όχι μόνο από τη Γαλλία μόνη της. Η ερώτηση που έχω και ίσως ε, η υποψία που έχω συχνά είναι αν όλα αυτά τα συμμερίζεστε. Νομίζω ότι καμιά φορά ε, υπάρχει φόβος για προηγούμενο, δημιουργία προηγουμένου και ότι ε, με αυτόν τον τρόπο θα βλάψουμε το ΝΑΤΟ. Για τα battle groups, για παράδειγμα, τις, ε, ομάδες, ε, τις μάχημες ομάδες. Αν θα μπορούσαμε να έχουμε άλλες δυνατότητες ή ας πούμε αν ε, στην περίπτωση του Μαλή ως Γερμανοί θα μπορούσαμε να έχουμε τρία τρανσάλ και να μεταφέρουμε μόνο Αφρικανούς και καθόλου Γάλλους. Πραγματικά όταν ε, διαβάζω ότι η κατάσταση είναι έτσι, αναρωτιέμαι τι θα γίνει την επόμενη φορά όταν έρθουν νέες απαιτήσει. θα έχει επιπτώσεις αυτό και στην γειτονιά μας ε, και στην εμπιστοσύνη που έχουν σε μας οι γειτονές μας. Πώς θα, βγούμε ε, από αυτή την περίεργη λογική. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας. Ήσασταν πολύ ρεαλιστικός η συνθήκη της Λισαβόνας μας έδωσε πολλά νομικά εργαλεία. Δυστυχώς, ενώ έχουν περάσει τα χρόνια, ε, δεν έχουμε σημειώσει αρκετή πρόοδο. Τα πράγματα είναι όπως, και ήταν, ε, όπως ήταν πριν από την ε, κύρωση της συνθήκης. Ελπίζουμε να έχουμε αρκετούς επαρκείς στρατιωτικούς πόρους, έτσι ώστε στο μέλλον να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Ε, φαντάζομαι ότι στο μέλλον θα έχουμε όλο και περισσότερους μικρούς εντό εισαγωγικών ε, πολέμους ε, και η Ένωση θα εμπλέκεται σε αυτούς όλο και περισσότερο. ποια είναι η γνώμη σας για την κρίση η οποία έκανε την άμυνα να τεθεί στο περιθώριο στην Ευρώπη. Εάν δούμε τους προϋπολογισμούς των διαφόρων κρατών μελών, βλέπουμε την μικρή σημασία που δίδεται στις αμυντικές δαπάνες. Ε, πώς μπορεί αυτό να διαρθρωθεί ε, με την, αυτή την έννοια του pooling and sharing. Ευχαριστώ. Ε, ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Κρόνμπεργκ εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε άλλωστε. Θα ήθελα να σας ζητήσω ε, να σχολιάσετε κάπως τα στρατεύματα μάχης ε, και ε, ποια είναι η διαφορετική ερμηνεία που δίνουν σε αυτά η ΕΠΑ ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς, ποια συνέργεια δημιουργείται μεταξύ αυτών. Ε, ομάδες μάχης θα έπρεπε να είχαν χρησιμοποιηθεί στο Κονγκό όπου είχαμε αυτές τις 20 τις επιθέσεις ή θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στο Μαλί σήμερα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλαμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στρατηγέ σας ευχαριστούμε για την προσέγγιση σας η οποία ήταν εξαιρετικά ε, ρεαλιστική ε, και μας έδωσε και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα σας. Αναφέρατε ότι χρησιμοποιούμε τους εθνικούς μας πόρους προετοιμαζόμενοι για συγκρούσεις του παρελθόντος, ενώ το pooling and sharing έχει περισσότερο να κάνει με τη βιτρίνα και όχι τόσο με την πραγματική πρόοδο. Τρεις είναι οι ερωτήσεις μου. Ποια είναι η άποψή σας για το Ευρωπαϊκό ε, Πυραυλικό Αμυντικό Σύστημα. Οι, Ευρω... Ηνωμένε Πολιτείες αποσύρονται όλο και περισσότερο από την Ευρώπη. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, πώς είναι η Ευρώπη προετοιμασμένη για μία ενδυνάμει για έναν ενδυνάμει ρωσικό εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί ενδυνάμει να βαίνει ε, αυξανόμενος. Το 2009 η Ρωσία έκανε ευρείες στρατιωτικές ασκήσεις, όπου ε, δοκιμαστικά μέσα στο πεδίο των ασκήσεων θα ήταν η θεωρητική ε, προσγείωση σε πολλο έδαφος. Έχετε λάβει υπόψη το ρωσικό στρατιωτικό δόγμα. Και τρίτη ερώτηση. Μιλήσατε για τις κυβερνοεπιθέσεις και την ε, ε, άμυνα σε αυτό το πεδίο και πιστεύετε ότι ε, ενδεχομένως ότι αυτά τα θέματα αντιμετωπίζονται καλύτερα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η κυρία Παναγιώτου. Παναγιώτοβα, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Τη βασίσατε άλλωστε στη μεγάλη σας εμπειρία. Λαμβάνοντας υπόψη τη νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ και την, την αναδιαργάνωση της ε, κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας, σίγουρα είναι η αθήρητη ανάγκη να αναδιαμορφώσουμε τη στρατηγική ασφάλειας που έχουμε σήμερα. Πόσο μάλλον που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 οι δύο οργανώσεις, το ΝΑΤΟ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δρούν στα ίδια επιχειρησιακά κέντρα και ανταποκρινόμενες και δύο στις ίδιες προκλήσεις. Θα πρέπει να έχουμε μια ευφυή προσέγγιση, έξυπνη προσέγγιση με βάση το pooling and sharing. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν έχω δύο ερωτήσει να σας θέσω. Πρώτον, θεωρείτε ότι η υιοθέτηση μιας λευκής βίβλου για τις αμυντικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελέσει μια πλατφόρμα ανάλυσης για την άμυνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πώς έχει αυτή τη στιγμή και ποιες προκλήσεις θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον ή είναι κάτι που θα βελτίωνε τη συνέργεια μεταξύ των ε, κρατών μελών που έχουν προσχωρήσει στις δύο αυτές οργανώσεις και ποια είναι η δυνατότητα άμυνας σε διμερές, πολυμερές και διεθνές επίπεδο. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι κάπως πιο προκλητική, αν θέλετε. Έχουμε μια οικουμενική αρχή, βάσει της οποίας το εκάστοτε εθνικό σύνταγμα το εγγυώνται οι ένοπλες δυνάμεις της εκάστοτε χώρες μετά τη συνθήκη της ε, ε, Λισαβόνας, γιατί την κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνας εγγυάται κυρίως, ο, εγγυώνται κυρίως οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άντριου Νταφ, παρακαλώ. Στρατηγέ, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα πολύ καλά από αυτά που είπατε. για το πού και ποιος θα πρέπει να έχει την ευρωπαϊκή ηγεσία από πολιτικής άποψης. Υπάρχει σαφώς ένα πρόβλημα με το ΝΑΤΟ που είναι βασικά, ε, βασικά δηλαδή υπάρχει ένα πολιτικό κενό εκεί, δεν υπάρχει εκεί πολιτική βάση και σίγουρα υπάρχει πρόβλημα εντός της Ένωσης λόγω της κατακαιρματισμένης φύσης ε, του συστήματος διακυβέρνησης της Ένωσης και του περιορισμένου βαθμού αρμοδιότητας που έχουμε σύμφωνα με τις συνθήκες. Μπορούμε βεβαίως να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Είμαστε πολύ ευφυείς και δημιουργικοί όταν πρόκειται για πειραματισμό νέων μορφών διακυβέρνησης. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να εστιάσετε περισσότερο τα προβλήματα της έλλειψης ευθύνη σε αυτά τα θέματα. Πιστεύετε ότι αν αυξηθούν οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Καταρχήν θα ήταν αυτό δυνατόν και δεύτερον αρκετό ώστε να γεμίσει αυτό το κενό. Ή πιστεύετε ότι μια ισχυρότερη και πιο τακτική παρουσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τώρα θα δριάσει το Δεκέμβριο ε, για πρώτη φορά για να ασχοληθεί με τη διάσταση ασφάλειας και άμυνας. Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έπρεπε να παίξει πιο προφανή, πιο διακεκριμένο και πιο τακτικό ρόλο στην θέσπιση στρατηγικής αλλά και στη λήψη αποφάσεων. στη Βόρεια Αφρική ίσως να χρειαστεί να ε, οργανώσουμε μια περίπλοκη μεγάλης κλίμακας και μακράς διαρκείας επιχείρηση πολιτικού και στρατιωτικού χαρακτήρα. Αν όντως αληθεύει αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε ακριβώς ποιος θα είναι επικεφαλής μιας τέτοιας επιχείρησης. Ευχαριστώ κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, με εξαιρετικό ενδιαφέρον άκουσα τις ε, παρατηρήσεις του στρατηγού Νάουμεν καθώς και τις, ε, ε, τις σημειώσεις, τις παραμέτρους που επεσήμανε ε, στη σχέση ανάμεσα στην ε, επιχειρησιακή δυνατότητα του ΝΑΤΟ και στο τμήμα που αφορά στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Το ίδιο άλλωστε έθεσε και ο κύριος Γκάλερ ε, δεν νομίζει ο στρατηγός ότι το κόστος, δηλαδή το μειωμένο κόστος μέσα από συνέργειες στην Ευρώπη θα μπορούσε να μας οδηγήσει ταχύτερα ε, σε μια κοινή πολιτική άμυνας. Όταν παραδείγματο χάρη ε, εξακολουθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε να παράγουν τάγκ σε μια γραμμή και η Ευρώπη σε 16 γραμμές. Το κόστος έχει τεράστια σημασία και θα μπορούσαν με τις συνέργειες και τη συνένωση δυνάμεων ερευνητικών να μειώσουν πάρα πολύ το κόστος, ιδιαίτερα για χώρες που βρίσκονται σε κρίση. Όπως παραδείγματος χάρη η δική μου χώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά βεβαίως δεν είναι ευχάριστα για τις χώρες που έχουν πολύ εξελιγμένη αμυντική βιομηχανία, αλλά το σύνολο της Ευρώπης βρίσκεται σε κρίση και θα έπρεπε να σκεφτούμε και το οικονομικό μέρος μιας τέτοιας προσπάθειας με την ίδια αποτελεσματικότητα. Οι Ευρωπαίοι ξοδεύουν ποσοστό κεφαλαίων σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι μεγαλύτερο από την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε ενιαία παρέμβαση για αμυντικούς σκοπούς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Merci Σας ευχαριστώ πολύ. Στρατηγέ μου, πολλές ερωτήσεις και διάφορες. Σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και με χαρά θα απαντήσω μία προς μία, αν μου επιτρέπετε. Εσείς, κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε στις αρχές για την θέση και τη στάση της χώρας μου. Θα πρέπει να πω ότι τα λέτε έξω από τα δόντια. Ανήκω σε αυτούς που στην Γερμανία πάντοτε τονίζουν όποτε μπορούν ότι η προϋπόθεση για μια ουσιαστική συμβουλή της Ευρώπης είναι η αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων και ε, θα πρέπει ε, πάντοτε και οι Γερμανοί να βρίσκονται ε, στο πλευρό των συμμάχων τους στο Μαλί. Είπα, για το Μαλί είπα σε μια γερμανική εφημερίδα την Παρασκευή ότι δεν αρκεί να στείλει δύο μεταγωγικά αεροπλάνα η Γερμανία στο Μαλί και απλώς να μεταφέρει αφρικανικές δυνάμεις δεν αρκεί αυτό. Και τολμώ να πω ότι αυτό είναι ένα ε, θέμα που πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζουμε. Ξέρετε φυσικά ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες μιας ε, ε, κυβέρνησης συνασπισμού. Πάντοτε πρέπει να φροντίζει να βρίσκει μια ισορροπία. Και όταν δυστυχώς η απόφαση πρέπει να λαμβάνετε τρεις μέρες πριν από τις εκλογές ε, στη Γερμανία, όπως και σε άλλες χώρες, είναι η πολιτική ιδιαίτερα προσεκτική. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχίσει. Εμείς ε, οι Γερμανοί πρέπει να αλλάξουμε τη στάση μας και έχω ε, ήδη πολλές φορές πει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει η Γερμανία να είναι αλληλέγγυα ακόμα και ε, σε περιπτώσεις ε, που υπάρχει κίνδυνος, ρίσκο. Ε, δεν θα πρέπει όλη η Ευρώπη να καταραίει από αυτό. Θα πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε όταν μας λένε οι γειτόνοι μας ότι δεν μπορείτε να κάθεστε στην άκρη, πρέπει να σταθείτε στο πλευρό μας. Πραγματικά, κοιτάξτε τι γίνεται στο Μαλί. Μια τρομοκρατική ζώνη στο Σαχέλ είναι κάτι που ήδη έχει αναφερθεί ξεκάθαρα από όλους τους Ευρωπαίους και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε. Δεν γίνεται οι Γερμανοί, επειδή στο παρελθόν είχαμε καταχρεστεί την στρατιωτική μας δύναμη πάντοτε να ε, είμαστε ελεύθεροι να μην χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις μας. Είμαστε σε μια συμμαχία και πρέπει να δρούμε μέσα σε αυτή. Σε όλη μου την πορεία πάντοτε έλεγα αυτά τα πράγματα και γι' αυτό είχα πάντοτε τόσους φίλους ε, πολιτικούς ε, που ε, χαιρόταν να πάνε στο ΝΑΤΟ και να παίζουν το ίδιο τραγούδι. Έχουν πολλά αλλάξει στη Γερμανία και πραγματικά και στην Ευρώπη και πρέπει πραγματικά να σας ζητήσω να το σκεφτείτε αυτό. Εδώ και 40 χρόνια θεωρείται ότι οι γερμανικές δυνάμεις δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιηθούν ξανά όπως ε, στο παρελθόν. Έχουμε μάθει καλά το μάθημα, αλλά με την επανένωση της ε, ε, Γερμανίας που πήραμε 18 εκατομμύρια. που τους φέραμε από το ένα άκρο στο άλλο με την τυπική γερμανική ε, μέθοδο, άνθρωποι οι οποίοι ε, υποστήριξαν ένα κομμουνιστικό καθεστώς για τόσα χρόνια, ε, να πρέπει τώρα να είναι ειρηνιστές της Ευρώπης, γενικά όλα αυτά να τα κάνουμε όλα μαζί, είναι πολύ δύσκολο να γίνει μέσα σε μια γενιά. Είναι πολύ γρήγορα για μας. πόσο δύσκολη ήταν η πρώτη ε, εμπλοκή της Γερμανίας ε, στην πρώην Ιουγκοσλαβία, ε, θα το θυμάστε. Το πρώτο γερμανικό πλοίο πήγε τότε στην Αδριατική και θυμάμαι πολύ καλά τι είχε γίνει. Δεν είχα μιλήσει για την τύχη του πλοίου. Ήταν κάποιος πολιτικός στην αντιπολίτευση τότε που ε, με είχε κατηγορήσει που έστειλα αυτό το πλοίο παρόλο που ήταν εντολή του Υπουργού μου. Τότε το 1991 έγιναν όλα αυτά. Και σήμερα στο Αφγανιστάν έχουμε Γερμανούς στρατιώτες ε, που μάχονται σε καθημερινή βάση και δεν είναι χειρότεροι από τους ε, συμμάχους μας. Έχουν πέσει τόσοι στρατιώτες στο Αφγανιστάν και εμείς παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας. Άρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πρέπει όμως να πάμε παραπέρα και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη δική σας υποστήριξη πρέπει πάντοτε να μας λέτε ότι είμαστε σε ευρωπαϊκό έδαφος και πρέπει όλοι να δρούμε από κοινού. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο ρόλος που πρέπει να παίζει η Γερμανία. Τώρα για τα βιομηχανικά ζητήματα που θέσατε, σας ε, ε, παραπέμπω στην ε, ομιλία του Υπουργού Άμυνας Πανέτα στο Λονδίνο την παρασμένη Παρασκευή. Είπε ξεκάθαρα ότι εμείς οι Αμερικανοί πρέπει να συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους. Πρέπει γιατί ο προϋπολογισμός άμυνας των ε, ΙΠΑ θα πρέπει να περικοπεί ε, κατά ένα τεράστιο ποσό σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πάνω από 400 εκατομμύρια. Οπότε, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και το βιομηχανικό κομμάτι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το είπα και στην εισαγωγή μου. Έχουμε την καλύτερη βιομηχανία ελικοπτέρων στον κόσμο στην Ευρώπη. Τώρα κοπεί είναι από τα καλύτερα. Αν έχουμε ένα μεσαίου, ε, μεσαίων βαρών, πούμε, ελικόπτερο, εδώ για την Ευρώπη και να συνεργαστούμε με τους ε, Αμερικανούς, να μην τους ζητήσουμε χρήματα τώρα για την ανάπτυξη αυτού του ελικόπτερου, αλλά μετά να πρέπει να αγοράσουν το ελικόπτερο. Τότε πραγματικά διασφαλίζουμε θέσεις εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα. Υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα στα οποία εμείς είμαστε ως Ευρωπαίοι καλοί ή και καλύτεροι από τους Αμερικανούς. Δεν μιλάμε μόνο για τα μαχητικά αεροπλάνα. Μπορούμε σε κάποια πράγματα να είμαστε περήφανοι. Και αυτό είναι μια πρόκληση για όλους. Θα πρέπει να δούμε πού είναι αδύναμη η Αμερική και εκεί ακριβώς να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε κάτι και να το προσφέρουμε στους Αμερικανούς. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας από τους δρόμους που μπορούμε να ακολουθήσουμε και έχουμε τη δυνατότητα αυτό. Και αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να αναπτύσσουμε πάντοτε, να προσπαθούμε πάντα να αναπτύξουμε κάτι στην Ευρώπη που έχει ήδη εδώ και καιρό ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι σπατάλη χρημάτων. Και δεν είναι αδίκως που στο τέλος μας είπαν ότι το European Defense Agency δεν έχει επικεντρωθεί στην, ε, στις ανάγκες της αγοράς. Η νανοτεχνολογία είναι ένα παράδειγμα. Τα ρομπότ είναι άλλο παράδειγμα. Αυτά τα όρια μεταξύ βιολογίας και ρομπότ είναι τόσα πράγματα που έχουν εφευρεθεί στο εργαστήριο, είναι ένα τεράστιο τομέα. Εκεί μπορεί η Ευρώπη να αναλάβει ένα ρόλο. Γιατί σε πολιτικό επίπεδο ήμασταν, θα έχει και εκεί επιπτώσεις. Ας πούμε, δεν θα υπήρχε ποτέ το Airbus αν δεν είχε γίνει το Τορνέιντο. Πρώτα για μαχητικά αεροπλάνα δημιουργήθηκε το σύστημά τους και μετά για την Airbus. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές δυνατότητες. Κύριε Γκάλερ, ε, αυτό το άγχος που αναφέρατε ότι μπορεί να προσβάλλουμε το ΝΑΤΟ, νομίζω δεν υπάρχει πια. Έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να συζητούμε με όλους ε, τους εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και αυτό το που πρότεινα το να έχουμε μια μονάδα από την ευρωπαϊκή πλευρά και μία από το ΝΑΤΟ που θα ε, συνεργάζονται είναι κάτι που ποτέ ε, που δεν εγείρει κάποιες επιφυλάξεις. Για το pooling και sharing, για το Transal ήδη απάντησα όπως είπα, είδατε για το pooling και sharing που αναφέρεται πριν τη συνένωση και την κοινή χρήση είναι, ένας, είναι η πρώτη ας πούμε οδός που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Δεν είναι η τελική λύση, είναι το πρώτο βήμα. Μετά από το pooling και το sharing πρέπει να σκεφτούμε τις επιπτώσεις. Σημαίνει ας πούμε ότι από κοινού χρησιμοποιούμε και συνενώνουμε και τις ε, δυνάμεις ε, για την εκπαίδευση ή για τη διοίκηση των δυνάμεων. Πώς θα γίνει η διοίκηση από κοινού σε εθνικό επίπεδο. Αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε και προς το παρόν υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα γιατί Έχουμε διαφορετικές μορφές εξοπλισμού. Ας πούμε τώρα, ε, τι γίνεται με τα ε, Άλλοι έχουν το Transalp, άλλοι το Hercules. Ε, πολλές φορές πρέπει να δαπανούμε διπλά χρήματα και για το ίδιο πράγμα, για τις συνέργειες. είναι μια δύναμη. Φυσικά υπάρχουν ε, τέτοιες δυνατότητες και η Ευρώπη φυσικά μπορεί σε κάποιους τομείς ε, να συνεισφέρει προσθετικά. Συμπληρωματικά όμως, όπως η κυρία Γιαννάκου είπε στο τέλος, να μην ε, θεωρείτε την συνέργεια ως ε, ένα κομμάτι, ε, ως μια στρατηγική στην οποία η Ευρώπη θα είναι για τη soft defense υπεύθυνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες για το hard defense. Δεν θα είχε μέλλον αυτό. Στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ έχω δει ότι μετράνε οι φωνές μόνο αυτών που θέλουν να αναλάβουν πλήρες ρίσκο και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Θα ήταν λάθος, κατά τη γνώμη μου. Εμείς οι Ευρωπαίοι στις σειράξεις ε, του κόσμου αυτού να μπορούμε να δρούμε μόνο οικονομικά, ενώ μπορούμε να έχουμε και άλλη συνδρομή και πάντα να είναι οι ΙΠΑ πρώτοι, πρώτες, παρόλο που έχουμε μεγαλύτερο ΑΕΠ από τους Αμερικάνους και να είναι πάντα αυτοί που θα κάνουν θα συμμετάσχουν σε αυτές τις ε, δράσεις με τόσα χρήματα, όπως έγινε ας πούμε στο Μαλί με 500 εκατομμύρια. Τώρα για την αντιπυραυλική ε, άμυνα στην Ευρώπη. Κύριε Κέλλαρ, νομίζω ότι για αυτό το θέμα πρέπει πραγματικά να βρεθεί μία λύση η οποία θα πηγαίνει πέρα από την Ευρώπη. Αποφασιστικό για την αντιπυραυλική άμυνα δεν είναι μόνο ποιοι είναι οι αντιπυραυλικοί μηχανισμοί που έχουμε και οι πύραυλοι, αλλά και ποιο είναι το σύστημα διαχείρισης μάχης που χρησιμοποιούν οι στρατιώτες με το οποίο συνδέονται δηλαδή τα όπλα τελικά. Όταν μιλάμε για πυράβλους πρέπει πάντοτε να γνωρίζουμε ότι μέσα σε 30 λεπτά μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ότι κάπου στον κόσμο εκτοξεύτηκε ένας πύραυλος. Πρέπει να το αυτοποιήσει λοιπόν κανείς προς τα που πηγαίνει ο πύραυλος και να βρει την αντίστοιχη άμυνα. Και αυτό πρέπει να το κάνει μέσα σε 15 λεπτά. Αυτό δεν μπορεί να περιοριστεί σε επίπεδο Ευρώπης. Στην αντιπυραυλική άμυνα, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια συνολική διαχείριση μάχης. Ε, μέσα από το ΝΑΤΟ, ας πούμε, ε, οι Αμερικάνοι αυτό κάνουν. Και μετά, σε επίπεδο μέσων άμυνας, μπορούμε να οργανωθούμε ευρωπαϊκά. Αλλά το σύστημα γενικά πρέπει να είναι παγκόσμιο. Αν σας κατάλαβα καλά, Είπατε επίσης ότι πρέπει να δράσουμε και στο επίπεδο του κινδύνου από τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία στρατιωτικά δεν είναι σε θέση, από τη στιγμή που η Ευρώπη είναι στο ΝΑΤΟ, να είναι επικίνδυνη για την Ευρώπη. Το κίνδυνος που βλέπω για την Ρωσία είναι ότι πολύ σύντομα μπορεί να χρησιμοποιούν ε, πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με τους Ρώσους. Και ένας ε, τέτοιος πόλεμος θα είναι κάτι που, είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε. Και γι' αυτό είναι σημαντικό η αποφασιστικότητα και η συνεργασία στο ΝΑΤΟ να δείξει στη Ρωσία ότι ε, δεν έχει καμία πιθανότητα να κάνει κάτι κατά της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ και ότι θα πρέπει να βρει τρόπους συνεργασίας έτσι ώστε να μπει μέσα στον δρόμο των διαπραγματεύσεων η επίλυση του θέματος ε, των πυρηνικών. Για το θέμα ε, του κυβερνοχώρου, κυβερνοπολέμου, πραγματικά είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Κάθε μέρα βλέπουμε τέτοιες επιθέσεις και σε επίπεδο άμυνας και εμπορίου. Οικονομικά τα κράτη επιβαρύνονται. Στην ΙΠΑ εκατοντάδες ε, χιλιάδες ε, δολάρια δίνονται για προστασία από αυτές τις επιθέσεις. Αυτό που υπόθηκε στην Ταϊβάν, αν το λάβουμε πραγματικά σοβαρά υπόψη, τότε η Κίνα προσπαθεί να φτιάξει ένα στρα... τρόπον την άστρατό που θα μπορεί ε, να κάνει κυβερνοπόλεμο και να σβήσει ε, σε επίπεδο ηλεκτρονικό μια ολόκληρη χώρα. Για πολλές μέρες. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της προστασίας από τον κυβερνοπόλεμο. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη στρατιωτική διάσταση, έχει να κάνει με τις συνολικές υποδομές ενός κράτους. Πρέπει να βρούμε μια ευρωπαϊκή λύση και μετά να τη συνδέσουμε ε, με μια διατλαντική λύση. Θα πρέπει λοιπόν να σας επιστήσω την προσοχή και να σκεφτείτε ότι αυτό δεν είναι απλώς το παιχνίδι κάποιων ε, hacker στο ίντερνετ. Υπάρχει πραγματικά θέμα και μπορεί πραγματικά να παραλύσει ένα ολόκληρο κράτος. Έρχομαι από τη χώρα του Κάλστον Κλάουσεβιτς. Ο Κλάουσεβιτς είπε κάποτε ότι σβήνει κανείς τον εχθρό του αν ε, του εξαλείψει όλα τα μέσα που διαθέτει. Τον 19ο αιώνα αυτό ήταν σωστό. Τώρα, στον 21ο αιώνα, σβήνει κανείς ένα κράτος αν μπορέσει να, το κάνει... να βοηθήσει στην παράλυση των ε, διοικητικών του μέσους, μέσων. Preventive παράλυση, λέγεται αυτό. Και αυτό το ξέρουμε και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Μιλήσατε, κύριε Βουλευτά, για ένα, μια λευκή βίβλο. Δεν θα ήταν παράλογο να είχαμε και μια λευκή βίβλο για τους Ευρωπαίους πολίτες, το οποίο θα λέει ότι δίνονται 200 εκατομμύρια ευρώ για την άμυνα στην Ευρώπη και τίποτα δεν επιτυχάνεται σε αυτό το επίπεδο. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων με έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο. Και σε αυτό το επίπεδο οι ευρωπαϊκές κοινέ ενόπλες δυνάμεις μπορεί να είναι πιστικές. Όταν σφίγγει τόσο πολύ το ζωνάρι, όλοι γινόμαστε πιο λογικοί. Ίσως με αυτόν τον τρόπο τελικά να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι. Τα εθνικά συντάγματα, αν το κατάλαβα σωστά, ε, είναι το καθήκον των ενόπλων δυνάμεων να ε, προστατεύει το Εθνικό Σύνταγμα. Όχι, είναι ε, καθήκον τους ε, να προστατεύουν τους ανθρώπους και την καιρότητα της χώρας. Το κατάλαβα σωστά, δεν ξέρω. Ίσως σε κάποια συγκεκριμένη χώρα να υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Δεν ξέρω αν το κατάλαβα σωστά. Ναι, Εάν κάνουμε τον παραλληλισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αναρωτιέται κανείς γιατί δεν έχουμε ευρωπαϊκό στρατό για να προστατεύει το ευρωπαϊκό μας σύνταγμα, που είναι δηλαδή η συνθήκη της Λισαβόνας. Ναι, ναι οπότε μάλλον δεν σας κατάλαβα καλά για το θέμα της πολιτικής διακυβέρνησης και της έλλειψης ευθύνης που αναφέρατε πριν, κύριε Βουλευτά. Νομίζω ότι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζει ε, τη διαχείριση κρίσεων. Χρειαζόμαστε στην πολιτική όλα τα εργαλεία. Και μια τέτοια χαμηλή σεντάσεως χρήση των ενόπλων δυνάμεων είναι καλή. Όμως η πολιτική άμυνας είναι στην αρμοδιότητα των κυβερνήσεων και για την ΚΕΠΑ. Το Συμβούλιο έχει μάλλον αποτιακό περιφερειακό ρόλο. Θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε αν πρέπει να αλλάξουμε ή να ενισχύσουμε αυτό το ρόλο. Στο μέλλον θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένας παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή μόνο αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα γρήγορα να δρά και να ζητά από την Κομισιόν να ε, χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της ε, Αλλά αυτά είναι όλα μελλοντικά σχέδια. Αν θέλουμε να πάμε προς την σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει κάπως να κινηθούμε σε συνεργασία με τους Αμερικανούς και να δούμε εάν στο μέλλον τελικά θα έρθει μια μέρα που ο πρόεδρος ε, της Κομισιόν και ο Αμερικάνος ε, πρόεδρος ε, θα μπορούν να συζητούν από κοινού και να λύνουν προβλήματα κρίσεων στον κόσμο. Είπαμε ότι στρέφονται οι Αμερικανοί προς την Ασία. Οι Αμερικάνοι χρειάζονται την Ευρώπη όμως. Είμαι ένας απλός ε, στρατιώτης και το μόνο που μπορώ να καταλάβω είναι ότι οι Αμερικάνοι είναι μια παγκόσμια δύναμη, αλλά για να παραμείνουν πρέπει να ε, έχουν και τη συνδρομή της άλλης όχθης. Χωρίς ε, τη συνδρομή της Ευρώπης και, και εμάς η δεν θα ήταν παγκόσμια δύναμη. Και εμείς Ευρωπαίοι θα πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να έχουμε σταθερότητα και ασφάλεια στην ε, απέναντι όχθη των Αμερικανών και να τους παρέχουμε τη βοήθειά μας τη χρειάζονται που τη χρειάζονται σίγουρα στο μέλλον σε διάφορες κρίσεις. Ελπίζω να απάντησα σε όλες σας τις ερωτήσεις. Ε, ναι, απαντήσατε πληρέστατα στρατηγέ μου. Καλύψατε όλες τις ερωτήσεις. Ίσως το ότι δεν είστε πλέον ε, εν ενεργεία ε, σας δίνει και μεγαλύτερη ευθερία να μιλάτε πιο ελεύθερα. Ο κύριος Λανσπέρκης ήθελε να προσθέσει μια ερώτηση. Έχουμε ακόμα 7-8 λεπτά πριν από την επόμενη συνεδρία. Ας ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Λαντσμπέργης. Μην μιλήσεις για 7-8 λεπτά, έτσι. Χωρίς μικρόφωνο, μιλητής. As NATO was built up and grew as επειδή το ΝΑΤΟ έχει δημιουργηθεί και μεγαλώσει ως Ευρωατλαντική Συμμαχία κατά διαφόρων ε, επιθέσεων, διαφόρων ειδών επιθέσεων, ε, είδαμε ότι πρόσφατα αλλάζει η κατάσταση αφού οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούνται ότι είναι πιο ισχυρό πυλώνα για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης και των χωρών της Βαλτικής από ό,τι φαίνεται όμως τώρα αλλάζει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή οι Αμερικανοί φαίνεται σαν να μας λένε να πηγαίνετε βρείτε και κατασκευάστε τους δικούς σας πυλώνες. Οι ΕΠΑ φαίνεται να συνεργάζονται με διάφορους άλλους και με διαφορετικούς τρόπους. Η Ευρώπη θα μπορέσει να σταθεί μόνη της, να σταθεί στα δικά της πόδια. τι σχετικές, τι σχετικές προβλέψεις υπάρχουν αφού η ευρωατλαντική μας ε, συμμαχία και ο στρατηγικός μας σχεδιασμός ε, στην ουσία ε, παρασύρεται από την πολυπαγκόσμια παγκοσμιοποίηση μάλλον υπάρχει κίνδυνος αν τέτοια παγκοσμιοποίηση καλύπτει ή στην ουσία ε, οδηγήσει σε μια νέα μορφή απομονωτισμού ή μια ευρωπαϊκή αδυναμία να μπορέσει να σταθεί, να δουλέψει στεναρά για μια ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα. Ευχαριστώ. Thank thank you very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πάλι γερμανικά. Έτσι μου είπανε τουλάχιστον να κάνω. Θα ήταν καλύτερα κάποιες φορές να μιλάμε ε, στα αγγλικά γιατί είναι λίγο πιο διφορούμενα και απαντάμε πιο εύκολα. Αλλά θα μιλήσω γερμανικά. Θα έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά με τα γαλλικά. Είμαστε πολύ πιο ε, ουσιαστική βέβαια εμείς ε, από ότι οι Γάλλοι. Αν σκέφτεστε την εποχή του ψυχρού πολέμου, τότε είναι λάθος να σκέφτεστε ότι μια αντιπαράθεση, η αντιπαράθεση ε, στον ψυχρό πόλεμο αποφασιζόταν στην Κεντρική Ευρώπη αποφασιζόταν στον Ατλαντικό. Από τη στιγμή που η ΕΠΑ δεν ε, θα ήταν σε θέση να ε, έχουν ισχυρή θέση, οι Ρώσοι θα είχαν κερδίσει. Το αποφασιστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ασφάλειας ήταν ο έλεγχος επί του Ατλαντικού. Και ίσως αυτό να ισχύει και για το μέλλον ακόμα περισσότερο. Αν δείτε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, τότε από το 2030 και μετά μπορεί να έχουμε έναν αρκτικό και παγωμένο με δραματικές συνέπειες για την ε, παγκόσμια οικονομία. Γιατί πραγματικά είμαστε εξαρτημένοι από ε, αυτόν σε επίπεδο εμπορικό. Θα μειωθούν οι πλωτές οδοί. Και ε, το πώς ελέγχουμε και παρακολουθούμε την κατάσταση και πώς θα γίνει αυτό στο μέλλον ακόμα δεν έχει ρυθμιστεί. Αν θα το κάνουμε εμείς ε, μόνοι ως Ευρωπαίοι δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε παρόλο που είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από αυτό. Ε, πρέπει να το κάνουμε ίσως σε συνεργασία με τη ΣΥΠΑ γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ακτών οι Ρώσοι το θεωρούν δικό τους. Ένα άλλο θέμα που αναφέρεται είναι ότι έχουμε κοινέ πεπιθήσεις και αξίες με τους Αμερικανούς. Εμείς οι Ευρωπαίοι με τους Αμερικανούς και τους ε, Καναδούς, ίσως και με τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς, έχουμε τα ίδια συστήματα κράτους δικαίου και δημοκρατίας. ένα δις από τους 7 με 8 δις ανθρώπους που ανήκουν σε αυτές τις χώρες στο μέλλον, που θα έχουμε στη γη στο μέλλον, ε, είναι πεπισμένοι για τη δημοκρατία και την ακολουθούν παρά τις αδυναμίες τους. Όμως ε, δεν αρκεί πάντοτε να προστρέχουμε στις αξίες και να τις επικαλούμαστε θα πρέπει να τις ε, προστατέψουμε. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για μένα. Γιατί ε, ουσιαστικά αυτό, αυτό μας σωθεί στο να διατηρήσουμε την ε, διατλαντική συμμαχία. Ένα τρένο πάντοτε πάνω σε δύο ράγες ε, τρέχει. Αν εμείς λοιπόν δεν έχουμε τη συνεισφορά μας, ε, δεν προχωράει το πράγμα. Εμείς ε, δώσαμε το πρωτοπύριο για την άμυνα της Αμερικής κατά τον ψυχρό πόλεμο. Πλέον δεν παίζουμε αυτόν τον ρόλο. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πώς ε, θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια ε, ως αντίπερα όχθη της Αμερικής. Δεν πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε μόνο τη Μεσόγειο, αλλά και την περιφέρεια της Ευρώπης. Να προσπιζόμαστε τα συμφέροντα της ε, Ευρώπης και αυτό να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε ε, υπερασπιζόμενοι και την ησυχία και την ε, ειρήνη στη Βόρειο Αφρική. Και πρέπει να δούμε και πώς θα διασφαλίσουμε την ε, σταθερότητα και την ασφάλεια και στην Αγγής Ανατολή. Πολύ λανθασμένα θεωρούν ότι εξαρτώνται οι Αμερικάνοι από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι λάθος δεν εισάγουν πλέον οι Αμερικάνοι από εκεί πετρέλαιο, μόνο οι Ευρωπαίοι. Και από το 2030 ακόμα και στο αέριο θα είναι ανεξάρτητοι οι Αμερικανοί. Θα εξάγουν γιατί χρησιμοποιούν νέες μεθόδους που εμείς στην Ευρώπη ακόμα δεν, γνωρί, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Άρα υπάρχουν στρατηγικά συμφέροντα και είμαστε ήδη στο 2013. Και πρέπει από τώρα να σκεφτούμε τι θα γίνει το 2020 το 2030. Γιατί ε, ο προκριματικός αγώνας μέχρι να έχουμε την πολιτική συνένεση και συμφωνία είναι σημαντικός. Πρέπει ήδη λοιπόν το 2013 να συζητάμε για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου, για αυτές τις απαντήσεις σας. Μας δώσατε πολλές διευκρινήσεις, παρουσιάσατε και παραθέσατε πολλές προοπτικές, μας δώσατε και συμβουλές Ελπίζω να ακολουθήσουμε όσο δεν τον περισσότερες. Σας ευχαριστούμε για τη μαρτυρία σας. Θα μας βοηθήσει σε όλη αυτή τη συζήτηση που θα διεξάγουμε καθ' όλη τη διάρκεια του 2013, ώστε το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2013, του Δεκεμβρίου, ε, να λειτουργήσει επικοδομητικά και να προσφέρει ε, λύσεις οι οποίες θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες, να δώσει απαντήσεις σε χρόνια ερωτήματα που έχουν να κάνουν και με τη συλλογική άμυνα, της Ευρώπης αλλά και με την άμυνα της κάθε χώρας. Αναφέρατε τις ε, στρατηγικές θέσεις και την εξέλιξη στη στρατηγική θέση π.χ. των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κάτι που έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και πέρσι ε, με, επί τη ευκαιρία της δημοσίευσης της ετήσιας έκθεσης για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Όλες αυτές οι τάσεις ε, οι οποίες διαγράφονταν τα προηγούμενα χρόνια τώρα είναι μια πραγματικότητα και θα πρέπει να ε, λάβουμε τα μέτρα μας και να κάνουμε τις απαραίτητες μεταστροφές σε όλα τα επίπεδα, το επιχειρησιακό, το θεσμικό, το οικονομικό κτλ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και ελπίζουμε να σας έχουμε και του χρόνου όπου θα μας κάνετε πάλι του χρόνου την επισκόπηση της κατάστασης έτσι όπως θα έχει διαμορφωθεί τότε. Ελπίζουμε ε, με πιο ε, θετικούς τόνους. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Έχουμε μαζί μας τον στρατηγό Πατρίκ de είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε αυτή την ακρόαση με την ιδιότητά του του Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαδέχθηκε το στρατηγό Σιρέν, ο οποίος μας είχε επισκεφθεί επανειλημμένος όπως θα θυμάστε. Η Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια νέα υπηρεσία ο στρατηγός Παλτεζά ήταν ο πρώτος πρόεδρος, μετά ο στρατηγός Σιρέν και τώρα είστε εσείς κύριε Ντεγουζιέ. Έχουμε τους 27 ε, ε, αρχηγούς των εθνικών επιτελείων. Είναι το ανώτατο στρατιωτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε. Θα ήθελα να διευκρινίσω ευθύ αμέσω το γεγονός ότι ο στρατηγός Πατρίκ Ντεγουζιέ είναι Γάλλος στρατηγός από τη Βουργουνδία μια πολύ σημαίνουσα προσωπικότητα στις ε, τάξεις των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, ωστόσο δεν παίρνει σήμερα το λόγο με την ιδιότητα του Γάλλου στρατηγού. Παίρνει σήμερα το λόγο με την ιδιότητα του Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον στρατηγό κύριο Γουμπί, ο οποίος είναι Γάλλος ε, στρατιωτικός, στρατηγός, εκπρόσωπος της χώρας του ε, στο ΝΑΤΟ και αλλού και αυτός δηλαδή, ο δεύτερος ομιλητής είναι αυτός που θα μας παρουσιάσει τη θέση της Γαλλίας ε, για την κατάσταση στο Μαλί. Έχουμε την αποστολή η οποία θα αναπτυχθεί επί τόπου, την, ε, το επιβεβαίωσε το Συμβούλιο την περασμένη Πέμπτη. Σίγουρα θα μας μιλήσετε για την αποστολή αυτή. Ωστόσο, ο στρατηγός Πατρίκου Γουζιέ δεν είναι επικεφαλής των γαλλικών στρατιωτικών ε, δράσεων και επιχειρήσεων στο Μαλί. Τόσο από την, ε, την ε, Ευρωπαϊκή Αποστολή Εκπαίδευσης, το EUTM Training Mission, δεν έχουμε Ευρωπαϊκή ε, Αποστολή στο Μαλί, μόνο Γαλλική και γι' αυτό ο δεύτερος ομιλητής θα μας μιλήσει για αυτά. Εσείς κύριε Γουσιέ, αγαπητέ στρατηγέ, θα μας μιλήσετε για τα ευρωπαϊκά θέματα, ε, π.χ. την επιχείρηση Αταλάντη ε, κατά της πειρατείας, η οποία στεύθηκε και έχει στεφθεί μέχρι αυτό το σημείο με απόλυτη επιτυχία. Μεταξύ άλλων, θα έχετε την ευχαίρεια βεβαίως, έχετε την ευχαίρεια, εάν το επιθυμείτε, να μας πείτε και για το γεγονός ότι η κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας έχει μπει στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα γίνει συζήτηση στο τέλος του 2013 το Δεκέμβριο στη Σύνοδο Κορυφής. Τι σημαίνει αυτό για τη Στρατιωτική Επιτροπή. Ε, στο δικό σας επίπεδο συνεδρίασης έχετε ξεκινήσει τη δουλειά για να τροφοδοτήσετε με τροφή προσκέψη την Σύνοδο Κορυφής. Βεβαίως έχετε την ευκαιρία να κινηθείτε όπως νομίζετε στην ομιλία σας. Εμείς ε, σίγουρα θα σας θέσουμε ερωτήσεις ε, για θέματα της, ε, επικαιρότητα. Έχουμε ερωτήσεις και για τα battle groups, τις μάχημες μονάδες. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι η πρώτη φορά που έχω την τιμή και τη χαρά να πάρω το λόγο, ε, να απευθύνομαι στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, διότι μου δώσατε την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας ε, τις σκέψεις μου. Διότι, ε, όντας εγώ στρατιωτικός, γνωρίζω πόσο προνομιούχος είμαι αυτή τη στιγμή που έχω την δυνατότητα να σας απευθύνω το λόγο. Λίγους μήνες μετά από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λίγους μήνες μετά που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως και στρατιωτικός σύμβουλος της είπα της εκπροσώπου της κυρίας Άστον. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας λοιπόν ε, τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις μου ε, σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι πολύ μεταβαλλόμενο και θα ήθελα να επιλέξω αυτό τον άξονα. Γύρω από αυτό θα στραφεί η ομιλία μου ε, και δεν θα περιγράψω τόσο τη θέση και το ρόλο της Στρατιωτικής Επιτροπής, διότι φαντάζομαι ότι τη γνωρίζετε αρκετά καλά. Σήμερα λοιπόν οι αναμνήσεις ε, πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος έχουν θολώσει και ευτυχώς ε, ο εχθρός δεν βρίσκεται καθόλου πρώτων ευρωπαϊκών πυλών. Ωστόσο η διεθνής κατάσταση παραμένει αρκετά τεταμένη, είναι απρόβλεπτη και έχουμε νέου πολιτικού κινδύνους ένα νέο διακύβευμα πολιτικό, οικονομικό, στρατηγικό και περιβαλλοντικό και γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Άλλωστε ο πρόεδρος Φαν Ρομπόη μας το υπενθύμησε στις 10 Δεκεμβρίου του 2012 επί τη ευκαιρία της ε, απονομής του βραβείου Νόμπελ ε, Ειρήνης στο Όσλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δήλωσε ότι ε, όλα αυτά έχουν λειτουργήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λειτουργήσει. Σήμερα η ειρήνη είναι κάτι το προφανές, ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο δεν σκεφτόμαστε καν, αλλά το ότι δεν το σκεφτόμαστε δεν σημαίνει σημαίνει ότι είναι και αδύνατο. Οι κοινωνίε μα δυσκολεύονται να καταλάβουν τη στρατιωτική δράση όταν αυτή λαμβάνει χώρα μακριά από αυτέ. Ε, ε, το ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε του κινδύνου με γυμνό μάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κιόλα. Η επικυρότητά μα μα το υπενθυμίζει διαρκώ. Μπορούμε να παραμείνουμε ε, αδρανεί όταν τρομοκρατικέ ομάδε απειλούν τι δημοκρατίε μα ή τη δημοκρατία φίλων χωρών. Μπορούμε να δεχθούμε όλε αυτέ τι επιθέσει πειρατεία ε, όταν ξέρουμε ποιο αντίκτυπο έχουν στην ασφάλεια του ανεφοδιασμού μας. Μπορούμε να δεχθούμε το κυβερνοέγκλημα ως ε, κάτι το μοιραίο από τη στιγμή που επιτίθενται ε, στα πιο ασφαλή μας δίκτυα. Σήμερα λοιπόν η αστάθεια της διεθνούς κατάστασης, η διαφοροποίηση των απειλών, το γεγονός ότι οι κρίσεις εμένουν και παραμένουν, ε, μας, κάνουν, μας οδηγούν σε ένα παράδοξο. Δεν έχουμε έναν συγκεκριμένο αντίπαλο αναγνωρισμένο με την παραδοσία και η έννοια του όρου, αλλά οφείλουμε να είμαστε συνέχεια σε επιφυλακή, κινητοποιημένοι και εκπαιδευμένοι για να υπερασπιστούμε τις αξίες μας αλλά και τα συμφέροντά μας. Οι απειλές του 21ου αιώνα είναι πολύ περίπλοκες, είναι διασυνοριακές και πολυδιάστατες. Ως εκ τούτου πιστεύω ακραδάντως ότι τις προκλήσεις ασφαλείας οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις συνολικά. Δεν μπορεί μια χώρα μόνη της μόνο. Πολλοί είναι οι διεθνείς παράγοντες που μπορούν να παρέμβουν στην διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι μία από τους μόνους παράγοντες, αν δεν είναι και ο μόνος, που μπορεί να κινητοποιήσει όλα τα σκέλη, και το πολιτικό σκέλος και το διπλωματικό και το οικονομικό και το νομικό και το αστυνομικό και το στρατιωτικό, προκειμένου να επιλύσει καλύτερα μία πολύ περίπλοκη κρίση και αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα ε, στο Σαχέλ. Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφαλείας και άμυνας είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Τα πρώτα θεμέλια τέθηκαν το 1999. Ωστόσο, το 2003 εγκαθιδρύθηκε αυτή η πολιτική με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας και την έναρξη των πρώτων στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων. Στον αιώνο μας ε, το γεγονός ότι τα μίντια ε, κάνουν τις εξελίξεις να επιταχύνονται και τις μεταδίδουν με τόσο ραγδαίο ρυθμό ε, αλλά και ενυπομονησία που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες δεν μας επιτρέπουν να καθυστερούμε και μειώνουν το βάθος του πεδίου στο οποίο παρεμβαίνουμε. Έχει γίνει μεταστροφή λοιπόν από πλευράς επιχειρησιακής, θεσμικής αλλά και από πλευράς δυναμικότητας, δυνατότητας της ευρωπαϊκής στρατηγικής δύναμης και τα, οι επιτυχίες ήταν, είναι απτές πλέον. Ως προς τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, οκτώ επιχειρήσεις έχουν ε, λάβει χώρα από το 2003. Για παράδειγμα, η επιχείρηση U4 στο Τσάντ έχει συμβάλει σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τον άμαχο πληθυσμό, για τους προσφύγες και τους εκτοπισμένους. Ήταν αυτή μια πολύ σημαντική διαφορά στο περιβάλλον ασφαλείας. Ήταν και η πιο ε, πολυεθνική στρατιωτική επιχείρηση που έχει λάβει ποτέ χώρα στην Αφρική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 14 κράτη-μέλη συμμετείχαν επί τόπου, 19 στο θέατρο των επιχειρήσεων και 22 στο αρχηγείο, στο στρατηγείο. Αλλά και η αποστολή εκπαίδευση ε, και κατάρτιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, ε, Σομαλία ήταν πολύ σημαντική. Εμβληματικό παράδειγμα ε, που δείχνει ότι οι αποστελέ μα πραγματικά κάνουν τη διαφορά επί τόπου. 3.000 στρατιώτες, αξιωματούχοι, αξιωματικοί που είχαν ήδη εκπαιδευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 550 στρατεύματα στο στρατόπεδο Μπιχάγκα τη Ουγγάντα που θα επιστρέψουν στο Μογκαντήσου στα τέλη Ιανουαρίου. Έχει δείξει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν αποστρέφεται του κινδύνου. Έδωσε την έγκριση στον επιχειρησιακό δεκητή τη επιχείρηση Αταλάντη να δράσει επί τόπου ε, ακόμα και σε χερσαία εδάφη όπου αυτό χρειαζόταν ώστε να εκπαιδευτεί ισχυρό μήνυμα στο κέρας της Αφρικής ε, και αλλάζοντας την αποστολή εκπαίδευση στη Σομαλία και κάνοντάς της να μπει σε διαφορετική φάση στο Μογκαντήσου με χάρη στην ε, επιχείρηση Αταλάντη και στις ευρωπαϊκές ναυτικές δυνάμεις οι πειρατείες στη Σομαλία είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, στο πιο χαμηλό δυνατό επίπεδο από το 2008. Οι πειρατικές επιθέσεις έχουν μειωθεί στις 35 φέτος συγκριτικά με τον αριθμό του, των 176 επιθέσεων το 2011 και θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε αυτή την εικόνα αναφέροντας την αποστολή εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαλί. Θα επανέλθω αργότερα σε αυτό. Όλες αυτές λοιπόν οι αποστολέ οι στρατιωτικέ και οι στρατιωτικές ε, καταδεικνύουν ξεκάθαρα την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει τη διαφορά στην επίλυση των κρίσεων και των συγκρούσεων. Ε, έχει σημειωθεί πρόοδος και σε, από πλευράς δυναμικότητας, δυνατοτήτων. Έχουμε στενή σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας, της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είμαι εγώ πρόεδρος, και του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, εγκαίρως όλα τα μέρη μπορούν να εμπλακούν, να συμμετάσχουν και να έχουμε ένα κοινό και ευρύ ε, μια κοινή και ευρία άποψη ε, για το ποιες είναι οι απαιτήσει ε, που θα χρειαστούν και που θα κληθούμε να παράσχουμε. Ε, πολλά κράτη-μέλη έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους ώστε να αποκτήσουμε ακόμα περισσότερες δυνατότητες, να αξιοποιήσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τους πόρους μας για να ξεπεράσουμε αυτό το κρίσιμο σημείο, για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Πολλά κράτη-μέλη λοιπόν έχουν δείξει την, τις έντονες φιλοδοξίες που έχουν σε αυτό το πεδίο, ενώ άλλα κράτη-μέλη είναι κάπως επιφυλακτικά δεν θέλουν τόσο να εκχωρήσουν εθνική κυριαρχία. Ε, θέλω να αναφέρω πιο συγκεκριμένα το European Air Transport Command, ε, το Ευρωπαϊκό αν θέλετε, Διοικητήριο Αερομεταφορών και εκεί συμμετέχουν ε, ε, στόλοι στρατιωτικών μεταφορών από τη Γερμανία, τις κάτω χώρες, το Βέλγιο και τη Γαλλία που έχει δείξει πόσο σημαντικό είναι τελευταία με τις τελευταίες εξελίξεις. Επίσης, η αμυντική συνεργασία στην οποία, την οποία έχουν εφαρμόσει οι σκανδιναβικές χώρες είναι ένα παράδειγμα συνεργασίας εξαιρετικά ενδιαφέρον και εξαιρετικά καινοτόμο, ειδικότερα ως προς την οργάνωση και την κατάρτιση. Ως προς την θαλάσσια εποπτεία, η πρωτοβουλία που έχει αναλυφθεί από 15 κράτη-μέλη με τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία μα επιτρέπει μια πολύτιμη ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών κυρίω ε, καλύπτοντα μεγάλο μέρο των ε, ευρωπαϊκών ακτών. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Όλοι έχουμε κοινά συμφέροντα και ενστερνιζόμαστε τι ίδιε αξίε. Θέλουμε να αυξήσουμε τη δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει τη διαφορά, όπου και να είναι παρούσα και όπου και να δρά. Ως προς τα πιο θεσμικά θέματα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δείχνει ε, πόσο ε, πόσες δυνατότητες έχουμε για να επιλύσουμε τα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Είναι το μόνο συντονιστικό όργανο που συγκεντρώνει και το ανθρωπιστικό σκέλος και το σκέλος για την ανακούφιση από τις φυσικές καταστροφές, ε, τις δυνατότητες διαχείρισης κρίσεων, την οικοδόμηση της ειρήνης αλλά και την ανεπτυξιακή συνεργασία. Συγκεντρώνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης όλες αυτές τις συνιστώσεις και μπορεί να δρά με πιο συντονισμένο τρόπο. Ως προς τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ε, επιτρέπει να μοιραζόμαστε πληροφορίες με όλες τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον επικεφαλής της Αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τους εκπροσώπους ε, των Ηνωμένων Εθνών. Στους κόλπους, στο πλαίσιο της Επιτροπής των Βρυξελών, του PSC και του CUMC. Ε, όλα αυτά δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μας ε, κάνει να ε, κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός ώστε η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαχείριση των κρίσεων να είναι ακόμα πιο αποτελεσματική. Σήμερα λοιπόν ο απολογισμός μας είναι αρκετά σημαντικός αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε γιατί η πρόοδος δεν είναι ανάλογη. Γνωρίζουμε ότι πολύ συχνά έχουμε χρηματοοικονομικούς περιορισμούς και γι' αυτό ορισμένα κράτη-μέλη μειώνουν σταδιακά αν όχι και ριζικά, τις πιστώσεις που δίνουν στο στρατιωτικό σκέλος των ε, προϋπολογισμών τους. Το παράδοξο σήμερα είναι ότι βλέπουμε μια Ευρώπη να αφοπλίζεται σε έναν κόσμο που όλο και περισσότερο εξοπλίζεται. Από το 2001 το σκέλος των στρατιωτικών δαπανών στην Ευρώπη μειώθηκε από το 29% στο 20%. Ε, ποια θέση θα έχει μια Ευρώπη 500 εκατομμυρίων ε, πολιτών εάν δεν διαθέτει ε, τις ικανότητες, τη δυνατότητα να εξασφαλίσει, να εγγυηθεί την ασφάλειά της. Αυτό είναι ένα δομικό ερώτημα, θεμελιώδες ερώτημα, διότι η φιλοδοξία φιλοδοξίες μας είναι αυτές που θα καθορίσουν και τα εργαλεία που τελικά θα επιλέξουμε, αλλά και αντιστρόφως τα εργαλεία που διαθέτουμε είναι αυτά που περιορίζουν ή πολλαπλασιάζουν τις φιλοδοξίες μας αναλόγως. Ο στρατογικός ε, απομονωτισμός σήμερα έχει τεθεί κατά μέρο. Πιστεύω ότι μόνο μία απάντηση προβάλλεται και είναι η εξή. Ε, πρέπει να έχουμε όλο και περισσότερη αλληλεγγύη, όλο και περισσότερες ανταλλαγές, όλο και περισσότερο μοίρασμα και κοινή συγκέντρωση, ούτω ώστε να αποφύγουμε ένα, ε, ένα διαρθρωτικό αφοπλισμό αν θέλετε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, σήμερα στρέφονται όλο και περισσότερο προ την περιοχή τη Ασία και του Ειρηνικού και μα ενθαρρύνουν προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε βεβαίω ούτε θέλουμε από του ιστορικού διατλαντικού δεσμού μα, ούτε εκείνοι το επιθυμούν. Μα καλούν όμω να εμπλακούμε όλο και περισσότερο ε, προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των συμπολιτών μα και να ε, συμβάλλουμε και εμεί στην οικοδόμηση τη ασφάλεια παντού. Και σε αυτή τη δυναμική εντάσσεται και η δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο κέρα τη Αφρική και στη Σαχάρα. Ε, θέλουμε να έχουμε μια ε, φιλόδοξη αλληλεγγύη, να μπορούμε εκ των προτέρων συλλογικά να προβλέπουμε τις εξελίξεις και να αναθεωρούμε και να εξετάζουμε συνεχώς το δυναμικό μας και τις ε, δυνατότητές μας. Υπ' αυτή την έννοια ε, θα πρέπει να έχουμε ασκήσεις και για να λαμβάνουμε σωστές αποφάσεις, να υπάρχει σωστή διάρθρωση και δομή της λήψης των αποφάσεων, για να μπορέσουμε να προβλέπουμε καλύτερα συλλογικά το τι μέλη γενέστε. Και θα πρέπει να εξελιχθεί και ο μηχανισμός ανάπτυξης ανάπτυξης όλου αυτού του στρατιωτικού δυναμικού, να συνεχίσουμε το pooling and sharing και να έχουμε καλύτερο συντονισμό. Η δημιουργία συγκεντρώσεων και συστάδων ε, στο χερσαίο επίπεδο, στο στρατιωτικό, το θαλάσσιο αλλά και το εναέριο σκέλος ε, θα μπορούσαν όλοι αυτοί να εξασκούνται και να κάνουν ασκήσεις με τον ίδιο τρόπο και θα μπορούσαμε έτσι να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την έννοια του pooling and sharing. Δεν είναι μόνο συμβολικό αυτό αυτές οι μονάδες ε, τις οποίες θα φτιάξουμε ε, αναλόγως με τις ανάγκες θα μπορούσαν να μοιράζονται και ιδέες ε, και στρατηγικά δόγματα αλλά και διαδικασίες εφαρμογής. Θα δείξουν και θα καταδείξουν ότι μπορούμε να έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόοδο στην πράξη χωρίς να θέσουν ένα αμφιβόλο, ένα την εθνική κυριαρχία που βεβαίως επιθυμούν τα κράτη και δικαίως να διατηρούν. Πάρα πολλά project αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και έτσι αυτά θα επιτρέψουν να αυξήσουμε τη διαλειτουργικότητα των στρατευμάτων μας τα επόμενα χρόνια. Ε, στο θέμα του π.χ. της αντιπυραυλικής βαλιστικής άμυνας, στο θέμα των μη επανδρομένων αεροσκάφων, στο θέμα του αποαέρος ανεφοδιασμού, ε, στις δυνατότητες αερομεταφορών, στο θέμα της στρατιωτικής, ε, της ιατρικής υποστήριξης των στρατιωτικών ε, επιχειρήσεων μπορούμε να, θέσουμε, να μοιραστούμε εργαστήρια, στρατιωτικά νοσοκομεία εκστρατεία. Όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα αναπτύξουμε από κοινού στα θέατρα των επιχειρήσεων. Και θα πρέπει να υπογραμμίσω και πόσο σημαντικό ρόλο ε, έχουν αυτές οι εργασίες πιστοποίησης και εναρμόνισης μέσα στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία για την πλοηγησιμότητα των στρατιωτικών αεροσκαφών. Έχουμε το φόρουμ ε, ΜΑΒΑ, για παράδειγμα Όλες αυτές οι προσπάθειες βελτιώνουν ε, την ε, διαλειτουργικότητα των στρατευμάτων μας. Και βεβαίως πιστεύω ακραδάντως ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις δράσεις ε, εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων στρατιωτικών μας. Ε, και πρέπει να γνωρίζουμε ότι για να αναπτύξουμε στρατιωτικές δυνατότητες χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο. Για παράδειγμα, για ένα άρμα μάχης από τη στιγμή που συλλαμβάνεται ως ιδέα μέχρι να αποσυναρμολογηθεί και το τελευταίο εξάρτημά του χρειάζεται να περάσουν 60 χρόνια. Για ένα πολεμικό σκάφος, πλοίο, ο χρόνος αυτός είναι 70 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέπουμε για να ε, ανταποκρινόμαστε σε όλες αυτές τις ε, πολιτικές. Είναι δύσκολο να προβλέπει κανείς το μέλλον. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι αν αρνείται κανείς να σκεφτεί το μέλλον και να προβλέψει τις αναταράξεις του, αυτό τον καταδικάζει να τις υποστεί τελικά. Θα ήθελα να επιμείνω στο γεγονός ότι το δυναμικό μας δεν μπορεί να, ε, να να, δεν, μπορεί να, δεν μπορούμε μόνο να το περιορίσουμε στο υλικό. Πρέπει να στρατολογήσουμε, να εκπαιδεύσουμε, να καταρτήσουμε το προσωπικό που χρησιμοποιεί όλο αυτό το υλικό και το προσωπικό είναι αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά σε, όλα αυτά τα, σε αυτό το πολύ απαιτητικό ε, περιβάλλον που, μέσα στο οποίο ζούμε και μέσα στο οποίο θα ζούμε σίγουρα και στο μέλλον. Ε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σίγουρα η, μια Ευρώπη άμυνα, ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο άμυνα είναι μια φιλοδοξία και εγώ θέλω να ε, ε, κάνω το παν για να συμβάλλω στην επίτευξη αυτού του στόχου στα τρία χρόνια της θητείας μου ως επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε διανύσει μια κάποια απόσταση. Η εδραίωση της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας μας επέτρεψε να σημειώσουμε πρόοδο σε θέματα ασφάλειας και άμυνας από το 2003 και μετά. Ωστόσο η πρόοδος αυτή είναι αρκετά εύθραυστη και θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι υπερεπτέρω. Ε, υπ' αυτή την έννοια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2013 θα εξετάσει όλα αυτά τα θέματα και με αυτή την προοπτική ε, στις 13 και 14 του περασμένου Δεκεμβρίου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάλεσαν την ύπατη αρμοστή, την ύπατη εκπρόσωπο, με συγχωρείτε, μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και μέσω της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσουν νέες προτάσεις για την ενίσχυση της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Το Δεκέμβριο του 2013 το ραντεβού είναι πολύ σημαντικό σημαντικό στη Σύνοδο Κορυφής δηλαδή του Δεκεμβρίου και εμείς θα πρέπει να επιδείξουμε ώστε να το μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Ε, εγώ είμαι αποφασισμένος να κάνω το παν για να συμβάλλω στην επιδίωξη αυτών των στόχων. Ε, θέλησα να μοιραστώ μαζί, μου, μαζί σας όλες αυτές τις πεπιθήσεις. Ελπίζω να μπόρεσα να σας περιγράψω τον οδικό χάρτη που θα ακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια του 2013 ε, και νομίζω ότι για περισσότερες λεπτομέρειες είναι καλύτερα να απαντήσω ξεχωριστά στις ερωτήσεις που τυχόν θα μου θέσετε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, στρατηγέ μου. Όντως, ήθελημένα επιλέξατε να μας παρουσιάσετε τη φιλοσοφία σας για τους επόμενους μήνες και νομίζω όντω πως είναι χρήσιμο να θυμίσουμε το στρατηγικό και πολιτικό αλλά και φιλοσοφικό πλαίσιο είναι αλήθεια των δράσεων που θα χρειαστεί να κάνετε στο πλαίσιο της ε, Στρατιωτική Επιτροπής. Τώρα εσείς ε, συγχωρήστε με γιατί εγώ θα σας προσγειώσω κάπως. Η ε, πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό θυμήσατε ότι είσαστε επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής, ότι από αυτή την ιδιότητα είστε σύμβουλος της ΥΠΑ της για τα στρατιωτικά ζητήματα. Μιλήσατε πολύ για πρόβλεψη στο ρόλο σας, στο ρόλο της Συντατικής Επιτροπής, στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβλέπει τις προκλήσεις και τις απειλές στο επίπεδο ασφάλειας. Επιτρέψτε μου να επανέλθω λοιπόν στην ε, επίκαιρη, στο επίκαιρο θέμα, το θέμα του Μαλή θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι εγώ εδώ κάπως έχω μπερδευτεί όσον αφορά την πρόβλεψη, γιατί είναι ένα ε, θέμα το οποίο δεν το ανακαλύπτουμε με την ε, Ισλαμιστική επίθεση της 10ης Ιανουαρίου είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό όπως και εσείς που μόλις αναλάβατε αυτές τις ευθύνες ε, με εκπλήσει το ότι εκπλαγήκαμε και όταν λέω εκπλαγήκαμε εννοώ όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι μόνο μια χώρα μπόρεσε να αντιμετωπίσει αυτή την, την έκπληξη η Γαλλία και με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι δεν υπήρξε μια πιο γρήγορη συλλογική απάντηση και κυρίως, και αν υπάρχει εσείς θα μου το πείτε, ε, ότι δεν είχε υπάρξει πρόβλεψη, σχεδιασμός για το τι θα μπορούσε και το τι θα να είναι και ποιοι θα ήταν οι κίνδυνοι και απειλές στο Μαλί, δεδομένου ότι είχαμε προβλέψει αυτή την ε, αποστολή, την EUTM, για την, ε, την κατάρτιση που προετοιμαζόταν, εντάξει επιταχύνθηκε τώρα, αλλά προετοιμαζόταν εδώ και πολύ, πολλούς μήνες. Και έπειτα ε, η ύπαρξη τρομοκρατών στο Μαλί ήταν κάτι που υπήρχε, ήταν γνωστό στη ε, Γενικά Επιτελεία και γι' αυτό με εκπλήσει η, η έκπληξη με την οποία έγινε ε, δεκτό, αυτή η επικαιρότητα. Και έπειτα μια γενικότερη ερώτηση που άμεσα συνδέεται με το Μαλί όμως, το θέμα της επέμβασης εκεί. Εσείς περιγράψατε όλη την προπαρασκευαστική εργασία, την πολύ μακρόπνοη που θα πρέπει να γίνεται για να αυξηθεί η διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών στρατιών. Εγώ να σας πω ναι, αύξηση της διαλειτουργικότητας, πολύ ευγενής στόχος, αλλά με είναι να μένουν με σταυρωμένα τα χέρια, ποιο είναι το νόημα όλων αυτών των προσπαθειών, των μακρόπνων, για ένα τόσο ισχνό αποτέλεσμα, όταν τελικά δηλαδή μόνο ένα στρατός πάει. Δεν χρειάζεται καν η διαλειτουργικότητα γιατί είναι μόνος του στο θέατρο των επιχειρήσεων. Εντάξει, θα μου πείτε ότι υπάρχει βοήθεια υλικό κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λίγα πράγματα Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην ενέργεια της προσπάθειας, τα λόγια επίσης ε, που έχουν ακουστεί για την προετοιμασία, για τη διαλειτουργικότητα, το σχεδιασμό και μετά στην πράξη το αποτέλεσμα είναι ισχνότατο σε σχέση με το τι θα μπορούσαν να είναι οι δυνατότητες των 27 συγκεντρωμένων. Είναι κάπως ευρύ το ερώτημά μου, ναι, το παραδέχομαι. Αλλά και κάτι πιο ε, χαρακτηριστικό ίσως, η Στρατιωτική Επιτροπή είπατε ότι την συναντήσατε πριν, λίγο πριν, είναι ένα τμήμα της απάντησης. Ήθελα να γνωρίζω λοιπόν αν από τις 10 Ιανουαρίου έχει συνεδριάσει η Στρατιωτική Επιτροπή για να μιλήσει για την κρίση του Μαλή. Ένα κράτος μέλος της Ένωσης είναι σε πόλεμο. Δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Συγκλήθηκε έκτατη συνεδρίαση της Στατικής Επιτροπής, όπως ε, έγινε εξάλλου και έκτατο ε, Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου λιγότεροι από τους μισού ήταν παρόντες, για να δείτε δηλαδή πόσο μεγάλη προτεραιότητα δίνουν. πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι δικό σας πρόβλημα. Αυτά ήταν οι ερωτήσεις μου. Ο κύριο Γκάλερ τώρα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Κύριε Στρατηγέ. Ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Λέτε ότι είναι η πρώτη σας φορά. Ελπίζω πιο συχνά να σας βλέπουμε στο εξή ε, και να φέρνετε πάντοτε καλά νέα. Θα ήθελα να συνεχίσω την ερώτηση του ε, συναδέλφου Ντανζόνα, στην οποία επέμεινε πολύ. Πραγματικά με εκπλήσει που τόσο εκπλαγήκαμε και σε επίπεδο Συμβουλίου δεν είχαμε ε, μια στρατηγική σε επίπεδο Συμβουλίου εδώ και δύο χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και δεύτερον, τα στρατιωτικά μας σχέδια τα τελευταία δύο χρόνια, κατά πόσον ε, συνδέονται με κάποια εμπλοκή στην περιοχή του Σαχέλ. Αν μιλάμε για ολοκληρωμένη προσέγγιση, ε, μιλάμε για πολιτικά, στρατιωτικά και αναπτυξιακά πολιτικά μέσα ταυτόχρονα. Πώς έχει κατάσταση τα τελευταία δύο χρόνια σε αυτό το επίπεδο. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Ιανουαρίου για μια ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή για συμβουλή στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μαλή. Στις 15 Οκτωβρίου ήδη είχε αποφασιστεί κάτι από ό,τι φαίνεται ότι ζητήθηκε ε, ο σχεδιασμός της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας ε, να επεκταθεί ως επίγον ζήτημα. Πέρασαν τόσοι μήνες από τότε. Δεν είχατε ήδη από τότε τη δυνατότητα για prudent planning, για την περίπτωση που κάτι μπορούσε να συμφωνηθεί. Από τις 15 ε, Οκτωβρίου μέχρι τον Γενάρη είναι τρεις μήνες. Και στο μεταξύ πήραν θάρρο οι εξτρεμιστέ ε, στο Μαλί λόγω της παθητικότητάς μας. Και πραγματικά ε, είναι πολύ λυπηρό αυτό. Και ε, αυτή την κριτική την είπα και στη δική μου κυβέρνηση. Γιατί δεν μπήκαμε ε, να συμμετάσχουμε ούτε στις εκπαιδευτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε και στις στρατιωτικές ε, ε, αποστολές, ούτε και στην μάχημη ομάδα, μονάδα. Εσείς πώς βλέπετε τη δυνατότητα μπλοκής της μάχημης μονάδας. Αυτή είναι η δική σας δουλειά. Εσείς προσφέρετε την ομάδα αυτή προς δράση. Ευχαριστούμε η κυρία Κόπα για τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας σε σχέση με το όραμά σας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Ωστόσο, βρισκόμαστε στα μέσα μιας πολύ σοβαρής οικονομικής κρίσης, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Μητική Βιομηχανία. Απόλυες θέσεις εργασίας, αλλά επίσης πολλά προβλήματα όσον αφορά τα, τις βιομηχανίες αυτές. Τώρα, για την κοινή έρευνα σε ορισμένα προγράμματα, σε αυτό το επίπεδο βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη περισσότερο προτιμούν να μοιράζονται παρά να συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους. Πιστεύετε πως ήταν ρεαλιστικό να συζητήσουμε για έναν πυλώνα της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά τις αποκλίνουσες απόψεις των κρατών μελών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Είναι βέβαια εξαιρετικά σημαντική κυριαρχία. Πώς βλέπετε εσείς τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, γιατί κατά τη γνώμη μου αντί να προχωράμε οπισθοχωρούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νικολάη. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ για το διορισμό σας. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Επιτροπή μας. Εντυπωσιάστηκα πολύ από την διάσκεψη για την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Ε, υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό που είπατε, ότι πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Μπορείτε να επεκταθείτε, είπατε think differently και έπειτα σε σχέση με τη συγκέντρωση και την κοινή χρήση δυνάμεων. Τι πιστεύετε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, κώδικας διοντολογίας, το πρόβλημα όμως είναι ο χρόνος όταν βλέπουμε την κρίση του Μαλή, νομίζω πως θα πρέπει να ελαφρυνθεί κάπως η διαδικασία, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τις αποφάσεις με εξαιρετικά γραφειοκρατικό τρόπο. Πώς ε, σκοπεύετε να επιταχύνετε τη λήψη απόφασης. Και τρίτη μου ερώτηση είναι φιλόδοξη, φιλόδοξη αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη υπάρχει ήδη ε, στη συνθήκη. Πώς μπορεί να γίνει πιο φιλόδοξη. Ευχαριστώ. Η κυρία Κρόνμπεργκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως βρίσκεστε σε μια μοναδική θέση για να κατανοήσετε πως τα κράτη-μέλη αντιλαμβάνονται την ανεξαρτησία και την κυριαρχία σε σχέση με την άμυνα τους. Και θα ήθελα να σας, γνωρίζ, να σας ρωτήσω ποιος είναι ο δικός σας ορισμός ανεξαρτησίας και κυριαρχίας ε, σήμερα στην Ευρώπη. Βλέπετε αλλαγές στην αντίληψη των κρατών μελών για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σαγκουράκης. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. εγώ είμαι από εκείνους που διαφωνώ κάθετα με τις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις στρατιωτικές, εκτός συνόρων. Και διαφωνώ με αυτές τις επιχειρήσεις γιατί θεωρώ ότι εξυπηρετούν συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών, την διασφάλιση των πηγών ενέργειας και πρώτων υλών και είναι σε βάρος των λαών. Δεν θα σας κουράσω με περισσότερες αναλύσεις, απλά θα σας θυμίσω κάτι που είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε. Ένας από τους τελευταίους προέδρους της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, απαντώντας γιατί υπάρχουν γερμανικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν, θεώρησε σκόπιμο να, να απαντήσει λέγοντας ότι εκεί που οι στρατιώτες ανοίγουν τον δρόμο πάνε μετά οι επιχειρηματίες. Ε, δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε αυξημένο βαθμό όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό το λόγο κιόλας η κατάσταση διεθνώς γίνεται όλο και πιο οξυμένη και πιο επικίνδυνη. Εξάλλου στην αναφορά σας το είπατε κιόλας. Είπατε δηλαδή επειδή οι Αμερικανοί πάνε στην Ασία, στρέψαν την προσοχή τους προς την Ασία, πρέπει, αν κατάλαβα καλά, να προσαρμοστούμε κι εμείς. Φυσικά οι Αμερικανοί πάνε προς την Ασία όχι λόγω τρομοκρατών, αλλά λόγω της ανόδου συγκεκριμένων κρατών εκεί πέρα όπως ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, ε, θέλω τη γνώμη σας για τα εξής δύο ζητήματα. Πρώτο ζήτημα, ε, έπεσε στην αντίληψή μου μια δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ της προάλλες όσον αφορά την υπερελιστική επέμβαση της Γαλλίας στο Μαλί, ότι το ΝΑΤΟ δεν θα ανακατευτεί στο Μαλί διότι δεν μπορεί να είναι παγκόσμιος χωροφύλακας. Και η ερώτηση μου είναι η εξής. Εάν στο Μαλί ο κίνδυνος των Ισλαμιστών τρομοκρατών όπως ονομάζονται και όπως λέγονται είναι τόσο μεγάλος το ΝΑΤΟ αδιαφορεί, το ΝΑΤΟ δεν το ενδιαφέρει, τι συμβαίνει. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και ότι βεβαίως υπάρχουν κίνδυνοι, αυτοί οι κίνδυνοι υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν, όχι όμως με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο για τον οποίο γινόμαστε μάρτυρες σήμερα. Δεύτερη γενική ερώτηση είναι η εξή: Επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της Σομαλίας, ειλικρινά Είσαστε ικανοποιημένο από την κατάσταση που ζουν οι Σομαλοί. Δηλαδή νομίζετε ότι με στρατιωτικές επιχειρήσεις τύπου σαν και αυτή που γίνεται στον, ε, στο κέρας Αφρικής με μια πολιτική των κανονιοφόρων, γιατί περί αυτού πρόκειται. Οι Σομαλοί θα δούνε άσπρη μέρα, όπως λέμε, θα μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματά τους και μου έκανε εντύπωση ότι δεν αναφερθήκατε σε αυτό. Και το λέω αυτό, ε, στρατηγέ μου, διότι δυστυχώς τέτοιου τύπου επιχειρήσεις είναι πάρα πολλές και ξέρετε, και στο Κονγκό έχουμε στρατιωτική παρουσία, αλλά και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αστάθεια, στρατιωτική αστάθεια. Έτσι δεν είναι. Αυτά διαβάζουμε. Τώρα ότι δεν μιλάμε για αυτά είναι επειδή είναι το Μαλί. Στο Νότιο Σουδάν που αποσχίστηκε από το Σουδάν στρατιωτική παρουσία θα έχουμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάει λέγοντας. Δεν σας ανησυχεί ότι όσο περνάει ο καιρός με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις διευρύνεται όλο και περισσότερο αυτό το τόξο τη ανασφάλεια, Merci beaucoup, Monsieur le Président. Σα ε, Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, στρατηγέ, για τις ευκρινήσεις ε, που δώσατε. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ μιας κοινή ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά αναφέρατε Άλλος υπηρεσίες ή οργανισμούς που ε, ασχολούνται με το τομέα της άμυνας. Ποιες είναι οι σχέσεις της Στρατηγικής Επιτροπής με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Merci. Bonne question. Σας ευχαριστώ. Ναι, η κυρία Γκόμες. Στρατηγία δεν μπόρεσα να σας ακούσω δυστυχώς, το, ε, το αναγνωρίζω γιατί βρισκόμουν ε, σε μια άλλη συνεδρίαση. Πολύ σημαντική. Ε, για τις επαφές με τις γυναίκες της νότιας όχθης της Μεσογείου είναι και αυτό πολύ σημαντικό θέμα και εκεί πρόκειται για θέμα αμήνη στην ουσία και ασφάλειας. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας δώσετε την άποψή σας για το πώς αυτή τη στιγμή η Ευρώπη άμυνας και ασφάλειας ενώπιον της γαλλικής ε, επέμβασης στο Μαλή, προστασία του λαού του Μαλί, ε, ασφάλεια κτλ. Αυτό το κάνουν ναι, για εκείνους αλλά και για μας. Η δική μας ασφάλεια απειλείται αν επιτρέπαμε να δημιουργηθεί εκεί ένα ένας ε, χώρος ε, προστασίας ε, τρομοκρατών αλλά και διαφόρων ειδών εγκληματιών. Ενώπιον λοιπόν αυτής της κατάστασης έχουμε τώρα βέβαια την, την τρομοκρατική επίθεση στην Αλγερία που πολλοί κατέκριναν την Αλγερία εννοώ ότι έδρασε βία ώστε να καταστήλει την τρομοκρατική αυτή ενέργεια. Αλλά φυσικά αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προκληθούν παρόμοια περιστατικά σε άλλες χώρες γειτονικέ στην περιοχή, όπως τη Λιβύη ας πούμε, που δεν έχει στρατιωτικές δυνάμεις τέτοιου τύπου. Και υπάρχουν όμως πολύ σημαντικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις για την ίδια τη χώρα αλλά και για την Δύση. Και όπου εργάζονται Ευρωπαίοι υπάλληλοι. Αυτό το εξετάζετε, στο επίπεδο, το εδεχόμενο το εξετάζετε στην Επιτροπή σας. Τα κράτη-μέλη προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν, να οργανωθούν, γιατί τότε η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει κάτι. Φυσικά σε συνεργασία με τις αρχές της Λιβύης, αν κάτι τέτοιο συμβεί στη Λιβύη. Και έτσι σκέφτηκα κι άλλη μια ερώτηση. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, της οποίας ηγείται η κυρία Άστον, θέτουν επιτάπητος θεμελιώδη ζητήματα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε κάθε είδους πρόκληση που δημιουργείται λόγω αυτής της κατάστασης. Ας πούμε, ένα μόνιμο γενικό επιτελείο ή θα δαπανούμε ε, τους πόρους ε, δεξιά και αριστερά. Μιλάνε για κοινή χρηματοδότηση επιχειρήσεων όπως αυτή του Μαλή. Γιατί εγώ Προέρχομαι από την Πορτογαλία και έχουμε θετικέ δυνάμει εξαιρετικά ικανέ να συμμετέχουν, αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν γιατί δεν έχουμε χρήματα. δεν θα πρέπει να δοθεί κοινοτική χρηματοδότηση, ή θα πούμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργό μα την περασμένη εβδομάδα, ότι δηλαδή ναι, πολύ θα θέλαμε, αλλά δεν έχουμε φράγκο. Τι στείλαμε, δύο, τρει, πέντε ανθρώπου, νομίζω. Το μήνυμο μου δηλαδή αν υπήρχε κοινοτική χρηματοδότηση θα μπορούσαμε ίσως να μοιραστούμε διαφόρων ειδών ε, δυνάμεις. Και τελευταία ερώτηση. Το ναυτικό. Κοινή πολιτική εν κοινοτική πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Τώρα είμαστε στο Μαλί. Δεν βρέχεται από τη θάλασσα η χώρα αυτή, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτό το είδους το πρόβλημα που έχουμε τώρα στο Μαλί θα μπορούσε να υπάρξει και σε πιο παραθαλάσσιες χώρες που είναι πολύ σημαντική περίπτωση υπόθεση θάλασσα. Για σκεφτείτε τον κόλπο της Γουινέας. Ξέρουμε ότι τη χρησιμοποιούν τα νότιο-αμερικανικά δίκτυα λαθρεμπόρων ναρκωτικών που μετέτρεψαν τη χώρα αυτή σε ε, κράτος ε, διακίνηση ναρκωτικών. Και από εκεί ξεκινά ένα σωρό προβλήματα, ξεκινούν ένα σωρό προβλήματα. Οριζόντια και κάθετα ε, δίκτυα έχουν δημιουργηθεί στη συνεργασία με τους Άραβες. Το ναυτικό λοιπόν περιλαμβάνεται, η συνεργασία των ε, ναυτικών δυνάμεων περιλαμβάνεται στα όσα κάνατε. Σα ευχαριστώ. Δεδομένου του χρόνου που έχουμε μαζί σας, ε, στρατηγέ, δηλαδή ένα τέταρτο και κάτι παραπάνω, δεν θα δεχτώ άλλε ερωτήσει, γιατί νομίζω πως έχετε ε, αρκετή δουλειά. Σα ευχαριστώ. Ναι, φανταζόμουν ότι θα μιλούσαμε λίγο για το μαλλί. Προφανώς. Εγώ τώρα τι μπορώ να σας πω για αυτό το θέμα. Φυσικά υπό την ευρωπαϊκή μου ιδιότητα και την ιδιότητά μου ως στρατιωτικού. Πάντοτε θα εκπλησώμεθα σήμερα όπως και αύριο και μεθαύριο από αυτές τις ε, χώρες. Η εισβολή του Σαντάμ Χουσέιν στο Κουβέιτ το σκεφτόμασταν, το είχαμε ε, ε, προβλέψει, αλλά παρόλα αυτά την ίδια εκείνη μέρα μας έπιασε εξαπρόπτου όταν πια έγινε. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για το Σαχέλ, για το Μαλί, ε, το, η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια είναι παρούσα σε αυτή την περιοχή του κόσμου και επενδύει σημαντικά ποσά για να σταθεροποιήσει, για να βοηθήσει αυτές τις χώρες. Και έπειτα προοδευτικά είχαμε μια εξέλιξη που ήταν καταρχήν μια εξέλιξη που οι ίδιοι οι κάτοικοι του Μαλή έπρεπε να αναλάβουν και να ανακτήσουν την ακαιρεότητα τον ε, της χώρας τους. Και με βάση αυτό είχε φτιαχτεί μια στρατηγική και αυτή η στρατηγική ακολουθήθηκε εδώ και χρόνια σε όλες τις εργασίες που έγιναν έτσι ώστε η αποστολή νουτή στο Μαλή να μπορέσει να αναπτυχθεί, να υπάρχει μια περιφερειακή ε, ιδιοποίηση, γιατί αυτό κάνει η υπηρεσία εξωτερική δράση. Χρησιμοποιεί το σύνολο των μέσων που έχει διαθέσει τη, ώστε να γίνει η ιδιοποίηση τη υπόθεση. Οι δυναμικέ δηλαδή που ε, λειτουργούν στην κάθε χώρα να αντιμετωπιστούν από τι ίδιε τι χώρε καταρχήν. Και αυτό γινόταν λοιπόν με την ε, στο Μαλί, αλλά είχαμε και την αφισμά, δηλαδή τις αφρικανικές χώρες, που στήριζαν. Όλα αυτά είχαν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και εκπλαγήκαμε. Όπως εξεπλάγει η διεθνή κοινότητα και από την εισβολή στο Κουβέιτ. Και έπειτα υπήρχαν δύο δρόμοι. Είτε επέμβαση του ΟΗΕ, επέμβαση μιας περιστασιακής συμμαχίας, επέμβαση μιας χώρας σόλο, αρχικά, ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μπορώ να σας πω ότι είτε πρόκειται για τους πρέσβεις, είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, είτε για τη δική μου επιτροπή, από την επαύριο της επέμβασης έγιναν ένα σωρό συνεδριάσεις ώστε να μοιραστούμε τις πληροφορίες και έτσι ώστε τα κρατημέλη, τα κρατημέλη που αποφασίζουν, να δούμε αν εντάσσονται ή όχι σε μια δυναμική. Δηλαδή, μια δυναμική που να είναι σε εξέλιξη σε σχέση με αυτό που είχε προβλεφθεί. Και αυτό κάναμε, επιτάχυνση δηλαδή τη ε, αποστολή για την εκπαίδευση των ε, ενόπλων δυνάμεων του Μαλιπού. Δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί ήταν απαραίτητο να εκπαιδευτεί μια, ένα στρατός, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει πόλεμος. Η απάντηση τη κυρία Άστον και τη εξωτερική υπηρεσία δράση και των κρατών μελών ήταν, ήταν σκόπιμο, γιατί οι απόψει και οι συμβουλέ που είχαν δοθεί ήταν ότι όντω πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος στρατός, νέο στρατός στο Μαλί και αυτό σήμαινε νέα, άλλου είδου συμπεριφορά, σεβασμό των πολιτικών αρχών και άλλου είδου συμπεριφορά επιτόπου, σύμμορφου προ τι δικέ μας αξίες. Ε, και γι' αυτό και η αποστολή μας αυτή στο Μαλί και ο στρατηγός Λεκουάντχα ε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μαλί και έρχεται αύριο, θα έρθει για να ε, ενημερώσει την ε, Στατιωτική Επιτροπή αλλά και τους πρέσβεις για το τι συμβαίνει στο Μαλί, να δούμε αν τα προγράμματα που έχουμε εμείς επεξεργαστεί ταιριάζουν ή πρέπει να τροποποιηθούν, έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια αποστολή που βασικό στόχο θα έχει να δημιουργηθεί ένας νέος στρατός στη χώρα αυτή, δηλαδή ε, κάτι αρκετά μακροπρόθεσμο. Όλα αυτά δείχνουν νομίζω ότι στο πλαίσιο των ε, ε, ευρωπαϊκών θεσμών δεν επικοινωνούμε αρκετά. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα διδάγματα που έχω αποκομίσει αυτούς τους δύο μήνες που έχω περάσει εδώ στις Βρυξέλλες. Ότι δηλαδή συμβαίνουν τρομερά πράγματα σε κάθε ένα από τα θεσμικά όργανα, αλλά τελικά δεν ε, γνωστοποιούνται. Εδώ στο Κοινοβούλιο ή και στο σύνολο του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Αυτό είναι βέβαιο. Και αυτό είναι ένας από τους στόχους που έχω. Δηλαδή, να γνωστοποιηθούν οι αξίες, οι δράσεις στις οποίες προβαίνουμε στο όνομα των κρατών από τους στρατιωτικούς που βρίσκονται όπου και αν βρίσκονται. Τώρα, διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών στρατών. Είναι κάτι το θετικό απαραίτητο, δεν κοστίζει πολύ. Είναι απαραίτητη η διαλειτουργικότητα γιατί αυτή μας επιτρέπει να γνωριζόμαστε καλύτερα και έπειτα ακόμα και διμερώς να μπορούμε να πέμβουμε όταν το επιθυμούμε και όχι απαραίτητο σε ένα ευρωπαϊκό συλλογικό πλαίσιο. Είναι λοιπόν απαραίτητο γιατί αυτό επιτρέπει ας πούμε, στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας εδώ και πολλά χρόνια να ε, κάνουμε κοινέ επιχειρήσεις όπου έχουμε σκάφη ε, με ελικόπτερα, με ε, ομάδες προστασίες μονάδες προστασίας ε, και κομάντο. Έχουμε περιπολικά αεροσκάφη του ναυτικού και κάθε, κάθε μια από αυτές τις μονάδες έχει δοθεί από διαφορετικό κράτος. Έτσι μπορούν λόγω χάρη της διαλειτουργικότητας να ε, συνεργάζονται με αποτελεσματικό τρόπο. Και δεν μπορούμε παρά να αναφέρομαι και την αποστολή εκπαίδευσης στρατιωτικών στην Σομαλία πάλι ε, και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν έχουμε το ίδιο πλαίσιο, το, την διαλειτουργικότητα δηλαδή. Από τις 10 Ιανουαρίου και μετά τι κάναμε. Δεν έχουμε σταματήσει, δεν έχουμε κάτσει ούτε λεπτό. Συγκαλούμε συνεδριάσεις, διαδίδουμε τις θέσεις των, των κρατών όσον αφορά τη... το Μαλί για να μπορέσουν να ληφθούν επίσημα οι αποφάσεις στην Στρατική Επιτροπή και μετά να παρουσιαστούν και στους πρέσβεις, ώστε να αποφασίσουν τα κράτη τι θα κάνουν. Και τώρα, επειδή είναι ο χρόνος λιγοστός, ε, την παρέμβαση των Battle Group, δηλαδή των μάχημων μονάδων, των τακτικών μονάδων ε, μάχης αυτές οι μονάδες έχουν ε, μια πρώτη βασική αρετή, δηλαδή διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα κράτη. Δημιουργείται διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα έθνη, τα οποία δεν είναι συνηθισμένα να έχουν ε, διαλειτουργικότητα. Διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή κοινοβουλευτικό, πολιτικό, διαρθρωτικό, Υπουργείο Αμήνης, Υπουργεία Αμήνη, Γενικά Επιτελεία Στρατού και έπειτα στο επίπεδο των μονάδων. Αλλά το βασικό δεν είναι οι μονάδε αυτέ. Είναι ολόκληρη η αλυσίδα αυτή για να μπορέσουν να λειτουργήσουν γρήγορα ε, εφόσον υπάρχει ε, μοιρασιά του βάρους θα πρέπει να υπάρχει εξ αρχής από το κοινοβουλευτικό επίπεδο να είναι προετοιμασμένοι ε, εκ των προτέρων. Και η δεύτερη αρετή αυτών των μονάδων, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν όλες είναι να μπορούν να επεμβαίνουν όταν συλλογικά θέλουμε να επέμβουμε. Δηλαδή, μια τακτική μονάδα μάχης είναι ένα εργαλείο, ένα εργαλείο όμως ενταγμένο σε πολιτικό επίπεδο. Μια τέτοια μονάδα δεν μπορεί να παρέμβει παρά μόνο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά έχει την πρόθεση να δεσμευθεί από πολιτικής και από στρατιωτικής άποψης. Δηλαδή, να διευθύνει την επιχείρηση αυτή μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιστεύω λοιπόν ότι το παράδειγμα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή που είναι το παράδειγμα του Σαχέλ και του Μαλή το εργαλείο δεν ήταν το κατάλληλο. Δεν ήταν το κατάλληλο ούτε από άποψη όγκους, όγκου, 2.000 άνθρωποι, δεν, όσον αφορά το πολιτικό πλαίσιο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι υπό κάποιες άλλες προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοιες ε, τακτικές μονάδες μάχης που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αλλά σίγουρα ε, λειτουργούν ως εργαλείο για να γνωριστούμε καλύτερα σε πολιτικό αλλά και στρατιωτικό επίπεδο ανάμεσα στα διάφορα κράτη. Σχεδιασμός. Αναφέρεται το χρονικά διάστημα προετοιμασίας ε, σχεδιασμού για να προετοιμαστεί δηλαδή μια εκπαιδευτική αποστολή. Η διάρκεια είναι η διάρκεια που θα πάρει η συνένεση ανάμεσα στα κράτη. Όλα τα κράτη δεν έχουν τις ίδιες γνώσεις για τις διάφορες περιοχές του κόσμου και αντιλαμβάνονται ότι από τη στιγμή που δεσμευόμαστε, δεσμευόμαστε σε μια μακροπρόθεσμη δυναμική, ότι αυτό είναι ένα από τα στοιχεία ανάμεσα σε άλλους όλων των τρόπων δράσης που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν διαπιστώνουμε ότι είναι θετική θετικό, αλλά φυσικά ε, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει και κίνδυνος και αυτός ο σχεδιασμός εδώ και κάποιες μέρες έχει επιταχυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εσείς μιλήσατε για τον βιομηχανικό πυλώνα αμήνης, βιομηχανία άμυνα. Εμείς δεν μπορούμε να την καθοδηγήσουμε τη βιομηχανία. Μπορούμε εμείς όμως στη στρατηγική να συμβάλλουμε από τη στιγμή που εκφράζουμε κοινέ ανάγκες ή που μοιραζόμαστε ένα όραμα για την προετοιμασία κοινού την κοινή προετοιμασία του μέλλοντος και πιστεύω ότι εδώ έχουμε πολύ πρόοδο ακόμα να κάνουμε ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες για αυτούς τους πυλώνες έτσι ώστε δηλαδή συλλογικά να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε καλύτερα το μέλλον και όχι να επηρεάσουμε ακριβώ, αλλά εν πάση περιπτώσει να είμαστε ένα ε, συνομιλητή πιο κατανοητό και πιο αξιόπιστο απέναντι στον βιομηχανικό ιστό, ο οποίο με τη σειρά του θα μπορέσει να οργανωθεί αντίστοιχα. Ε, εδώ η, υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αμήνη κάνει εξαιρετική δουλειά όσον αφορά την δικτύωση των διαφορών φορέων, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκέ χώρε να μπορέσουν, αν όχι όλοι μαζί, αλλά σε ομάδες, να μπορούν να έχουν μια κοινή οπτική, ένα κοινό όραμα. Πιστεύω πως μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς οι στρατιωτικοί στην έκφραση των αναγκών μας εάν ε, τις ανάγκες αυτές τις ε, γνωστοποιήσουμε στην βιομηχανία για το pooling and sharing την ε, συγκέντρωση και κοινή χρήση δυνάμεων. Πιστεύω πως είναι απαραίτητο αλλά δεν είναι καμία θαυματουργή λύση. Ε, δεν είναι θαυματουργή λύση γιατί άμεσα αναφέρε, ε, ε, προσκρούμε στα προβλήματα κυριαρχίας των κρατών, δηλαδή την εγγύηση πρόσβαση στις στρατιωτικές τους δυνατότητες. Και εγώ ως εκπρόσωπος του διοικητού του γενικού μας επιτελείου θα πρέπει να σας πω ότι προσέχει πάρα πολύ τις δυνατότητες ε, που μπορεί να τεθούν σε κοινή χρήση ε, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να μοιραστεί όπως ας πούμε τις επιθετικές μας ε, δυνατότητες αλλά υπάρχουν και άλλες που επίσης εξίσου δύσκολα μπορεί κανείς να μοιραστεί. Έχουμε ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα παράδειγμα με το, την Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Αερομεταφορών ε, προσπαθούμε να βρούμε επιλογές που θα επιτρέψουν ε, την κοινή χρήση σε άλλους τομείς. Αυτές οι συνεργασίες που κάνουμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μάλιστα του Δεκεμβρίου θα συζητηθεί αυτό, υπάρχουν επιλογές όσον αφορά την διοικητική στήριξη, τις τηλεπικοινωνίες, την δικτύωση, τα ξαποστάσους ε, ε, μάλλον πλοηγούμενα αεροσκάφη και ε, τις δυνατότητες να εξοικονομήσουμε σημαντικά ποσά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεών μας και όσον αφορά κυρίως τη δημιουργία συνέργειας ανάμεσα σε όλους μας. Ανεξαρτησία ή κυριαρχία στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ ιδιαίτερα πολιτικής φύσης βεβαίως, για το οποίο δεν έχω πολλά να πω, εκτός από την ελεξάρτηση. Εμείς ε, πρέπει να δημιουργήσουμε την αλεξάρτηση για τις νέες γενιές και βλέπω και χαιρετίζω εδώ νέους ε, Ικάρους, Γάλλους Ικάρους, ε, μου θυμίζει τα νιάτα μου να σας βλέπω εδώ ε, υπάρχει το σχέδιο Έρασμος που δεν έχει να κάνει με το στρατό, είναι το Έρασμος για τους στρατιωτικούς, δηλαδή ε, ανταλλαγή διαφόρων αξιωματικών, νέων αξιωματικών ανάμεσα στα κράτη. Έχουμε δηλαδή τομείς ε, που πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την ε, σε που θα δημιουργήσουν την αλληλεξάρτηση που είναι θετική ε, και αφήνει ωστόσο το κάθε κράτος ελεύθερο να μπορεί να προβαίνει στις επιλογές του. Δεσμεύσει τώρα και επεμβάσει εκτό των ευρωπαϊκών συνόρων. Εγώ θα αντιστρέψω την ερώτησή σα και θα επιμείνω σε ένα από τα σχέδια, ένα από τα θέματα που χρειάζεται να εξετάσω κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου, δηλαδή ε, η δέσμευση των στατικών εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, αλλά πρόκειται για την ε, ρήτρα της αλληλεγγύης. Η ρήτρα της αλληλεγγύης που δεν είναι η ρήτρα της κοινή άμυνας. Η ρήτρα αλληλεγγύης, όπως γνωρίζετε καλά, είναι αυτή που οδηγεί σε περίπτωση μιας μεγάλης τρομοκρατικής επίθεσης ή ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, για παράδειγμα, ε, κάποιο γεγονός που να οδηγούν ότι, στο γεγονός ότι οι, οι δυνατότητες του κάποιου κράτους ξεπερνιόνται και χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια από τα άλλα κράτη και να δεσμεύσει ακόμα και στρατιωτικά μέσα. Εδώ πρέπει να το σκεφτούμε, πρέπει να σχεδιάσουμε και να λύσουμε όχι τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσουμε επιτόπου, γιατί η δράση επιτόπου γίνεται αποτελεσματικά, γιατί θα είναι αποτέλεσμα επενδύσεων από κάθε κράτος, αλλά όσον αφορά το συντονισμό. Αν αύριο Έχουμε ένα Τσερνομπίλ στην Ευρώπη. Πώς θα ενεργήσουμε για να καθησυχάσουμε τον κόσμο χρησιμοποιώντας το σύνολο των δυνατοτήτων καταπολέμησης, ε, ανα, ανάλυσης ε, ε, και ανάσχεση των βιολογικών, χημικών και πυρηνικών όπλων. Έχουμε δηλαδή δουλειά να κάνουμε. Πρέπει να προβλέψουμε το απρόβλεπτο. Ε, αυτό θα μας επιτρέψει, ίσως όχι σε επιστατικό επίπεδο, αλλά τουλάχιστον στους κύκλους λήψης απόφασης, στους κύκλους του συντονισμού, να γνωρίζουμε καλύτερα τις δυνατότητες των άλλων, ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε πιο αποτελεσματικά τη στιγμή που θα υπάρξει ανάγκη. La relation du, du comité militaire avec... Euh, η σχέση της ε, στατική Επιτροπής με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αμήνης είναι φυσικά εξαίρετη και απαραίτητη, διότι η αρχηγοί των επιτελείων είναι αυτοί οι οποίοι ε, έχουν τα μέσα και άρα και την εμπειρία. Άρα πρέπει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Μήνες να είναι ο φορέας που θα επιτρέπει να, να, να, να υπάρξουν προσανατολισμοί όπου από κοινού ίσως θα πρέπει να υπάρξει έρευνα για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε έναν ε, κατάλληλο βιομηχανικό ιστό είτε για να αναπτυχθούν οι δυνατότητες που, που, που είναι απαραίτητες. Στον τομέα του διαστήματος έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας οι σχέσεις με το διάστημα είναι απαραίτητο τομέα για το στρατό, για να γνωρίζει, για να γνωστοποιεί, να επικοινωνεί και για να δρά, να ενεργεί. Μια μέρα χωρίς το διάστημα θα ήταν καταστροφή για όλους, για το οικονομικό σύστημα, για το τροπεζικό σύστημα και καταστροφή για τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις. Οι στρατιωτικές μας επιχειρήσεις εξαρτώνται πολύ από το διάστημα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εντατικοποιήσουμε την, ε, τη διάδραση με το σύνολο των ε, φορέων που δρούν στο διάστημα. Πιστεύω πολύ σε ένα τομέα που είναι η εποπτεία όχι από το διάστημα αλλά προς το διάστημα. Αυτό εξυπηρετεί ένα σκοπό, δηλαδή να γνωρίζουμε τι υπάρχει εκεί, να αποφύγουμε τη συνδετικοποίηση του διαστήματος, να επιτρέψει την εγγυήση των ε, ε, της πρόσβασης στο διάστημα από τους Ευρωπαίους ε, που, που έχουν αυτές τις δυνατότητες και να υπάρχουν και επαρκείς δορυφόροι. Ε, δορυφόροι αλλά και συνεργασία για να αποφεύγουμε τα τα σκουπίδια του διαστήματος. Μιλήσατε τώρα επίσης για ένα μόνιμο γενικό επιτελείο. Εγώ δεν μπορώ ανάποδα την ερώτηση, δηλαδή να πω τι χρειαζόμαστε, τι μας λείπει. Τι λείπει στους θετικούς, τι λείπει από την κυρία Άστον για να μπορεί καλύτερα να κάνει τη δουλειά της. Όσον αφορά την πρόβλεψη αλλά και την παρακολούθηση. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει τεράστιος δυναμισμός στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Είμαι δύο μήνες εδώ, είδα έξι μονάδες κρίσης, όπου συμμετείχαν ένα σωρό κόσμος, αντιπροσωπείες των ΟΗΕ, αντιπροσωπείες εδώ στις Βρυξέλλες, δηλαδή ε, πολλοί, πολλές επαφές που επιτρέπουν να γνωρίζουμε καλύτερα και να προβαίνουμε σε επιλογές. Μόνο που όταν ε, γίνουν οι επιλογές, ο σχεδιασμός περιπλέκεται, διότι δεν υπάρχει μόνιμη δομή σχεδιασμού που να αποτελείται από πολιτικούς και από, από το τμήμα το πολιτικό και το τμήμα το στρατητικό ώστε να ε, μπορούμε να εξετάσουμε τις διάφορες πτυχές. Συρία, ας πούμε, την επόμενη μέρα τι κάνουμε. Κάνουμε σχετικές εργασίες, αλλά δεν μπαίνουμε στις λεπτομέρειες όπως θα μπορούσε να κάνει ένας μόνιμος, μια μόνιμη δομή σχεδιασμού. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν θα έπρεπε να υπάρχει ένας, μια δομή παρακολούθησης, ε, ίσως κάποιος σχεδιασμός, ναι, να είναι απαραίτητος. Και φτιάχνεται, δημιουργείται σιγά σιγά. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι μόλις δύο ετών και είμαι βέβαιος ότι αν και συνεχίζοντας θα καταλάβει όλο για ένα και περισσότερο τις ανάγκες της. Γιατί φυσικά αυτό το είδος η δομή ε, παίρνει χρόνο για να οργανωθεί. Αν μπορώ να συνεχίσω, μπορώ να κλείσω ε, με το ναυτικό σκέλος της ε, πολιτικής αμήνας και ασφάλειας. Πιστεύω πως η επιχείρηση στα νησιά της Ομαλίας έχει επιτρέψει πολλά πράγματα για την Αφρική. Και για μας τους Ευρωπαίους ε, επέτρεψε να υπάρχει ασφάλεια για την ανθρωπιστική βοήθεια, για τις δικές μας, ε, το δικό μας ανεφοδιασμό, αλλά και έτσι, αν τα κράτη το θέλουν, ε, ομαδικά ή και διμερώς, θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις ναυτικές τους δυνάμεις για να εγγυηθούν το σεβασμό των, των θαλάσσιων συνόρων μας, τον σεβασμό του θαλασσίου περιβάλλοντός μας και νομίζω πως αυτό είναι καλό για το μέλλον, διότι οι εξελίξεις στον κόσμο το οδηγήσουν όχι σε ναυτικοποίηση, γιατί κάποιοι το χρησιμοποιούν πολύ αυτόν τον όρο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα καταστήσουν απαραίτητη την παρουσία μας στη θάλασσα όσο γίνεται περισσότερο, για να αποφευχθούν τα παράνομα εμπόρια, τα λαθρεμπόρια, αλλά και οι επιθέσεις ε, στον ναυτικό, ε, στους στόλου μας ή και στις παράκτιες μας, στα παράκτια μας συμφέροντα. Κοινή χρηματοδότηση τώρα, ε, να σας πω ότι εδώ επανέρχεται αυτή η συζήτηση, δεν υπάρχει λύση. Τα κρατη μάλλη δεν θέλουν να πάνε προς χρηματοδότηση, διότι βλέπουν απώλειες. Απώλειες αυτονομίας. Και άρα αυτό οδηγεί, εφόσον υπάρχουν ε, επεμβάσεις, να υπάρχουν δισταγμοί, ιδιαίτερα σε φάσεις κρίσης. Γίνονται προσαρμογές. Νομίζω πως αυτό είναι αναπόφευκτο θα πρέπει να πάμε πιο μακριά. Δεν ξέρω, υπάρχουν τομείς που θα έπρεπε να προχωρήσουμε περισσότερο. Αλλά πιστεύω πως είναι αρκετά παράλογο να έχουμε μέσα που να είναι σε έτοιμα, σε επιφυλακή. Σε ορισμένες χώρες υπάρχει προσωπικό ειδικό για αυτές τις ομάδες, τις μάχημες και έπειτα να μην λαμβάνεται υπόψη η χρηματοδότηση από το σύνολο από τη στιγμή που ε, επεμβαίνουν στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε βάση περιπτώσει, νομίζω θα πρέπει να επιμείνουμε και σταδιακά, αν δούμε, στο... αν δούμε το παρελθόν, εδώ και 5-6 χρόνια έχουν υπάρξει εξελίξεις. Νομίζω πως και εδώ είμαστε στον καλό δρόμο. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου. Νομίζω ότι αναφερθήκατε σε πολλά και διαφορετικά θέματα για πρώτη φορά είναι ήδη πάρα πολύ αυτό. Την επόμενη φορά θα μας επισκεφθείτε, σίγουρα θα εμβαθύνουμε περισσότερο σε κάποια από αυτά τα σημεία. Σε κάθε περίπτωση ελπίζω οι επαφές μας να είναι συχνές, αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός μας. Στόχος σας άλλωστε είναι να διαδώσετε περισσότερο την πληροφόρηση για τα τεκτενόμενα ε, σε εμάς εμείς ε, θέλουμε να σας πούμε ότι είστε πάντοτε ευπρόσδεκτος. Θέλω να εκφράσω την ελπίδα ότι γρήγορα θα απαντηθούν τα ερωτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοι. Σίγουρα οι δράσεις σε αυτό το τομέα εκτείνονται σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Ωστόσο, ε, πάντοτε καλούμεθα να ε, δράσουμε κατεπηγόντως, αναλόγως με τις εξελίξεις. Αυτό άλλωστε ε, απαιτούν και οι συμπολίτες μας και θα έλεγα ότι οι πολίτες πολύ συχνά φοβούνται και δεν καταλαβαίνουν καθόλου αυτή την χρονική διαφορά, τη χρονική καθυστέρηση που υπάρχει μεταξύ των εργασιών και των επιτευγμάτων μας ε, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των επιτυχιών ε, και του μεγέθους ε, αυτών των επιτυχιών επιτόπου στις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις. Μας βοηθήσατε λοιπόν να καταλάβουμε καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και για τις απαντήσεις σας και για την ε, παρουσίασή σας. Θα έχουμε λοιπόν τώρα ε, δύο λεπτά διάλειμμα περιμένοντας τον στρατηγό κύριο Ρουμπί. Θα συμπροεδρεύσω μαζί με τον κύριο Γιάν Πασκού γιατί είναι μια κοινή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για την Ασφάλεια και την Άμυνα και της Επιτροπής για τις Εξωτερικές Υποθέσεις.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

This is pulling and sharing. um, this was an example of pulling and Είδατε μόλις ένα παράδειγμα του pooling and sharing, της κοινής συγκέντρωσης πόρων και δυνάμεων. Αγαπητοί φίλοι, εκ μέρου τη Υποεπιτροπή για την Ασφάλεια και την Άμυνα και εκ μέρου τη Επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων, με χαρά ε, καλωσορίζω ε, τον Ζιλ Ρουμπί, που είναι ο στρατιωτικό εκπρόσωπο τη Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Ο Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, κ. Λογόν Φαμπιού, δεν μπόρεσε να έρθει τη Δευτέρα, που υποτίθεται ότι θα ήταν εδώ. Σε κάθε περίπτωση όμως η κατάσταση στο Μαλή είναι εξαιρετικά σημαντική και η γαλλική οπτική της κατάστασης είναι ακόμα πιο σημαντική. Αύριο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι θα, έχουμε, θα συνεδριάσουμε στις 9.30 και θα έχουμε άλλους ανώτατους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και με την απόψενή μας συζήτηση αλλά και με την αυριανή συζήτηση ε, ελπίζουμε ότι θα αποκομίσουμε μια περισσότερες γνώσεις για το τι συμβαίνει ακριβώς στο Μαλί. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα θυμάστε το μήνυμα αλληλεγγύης που εκπέμψαμε ε, προς τους Γάλλους φίλους μας ως προς την ε, γαλλική παρέμβαση η οποία ε, έλαβε χώρα ανταποκρινόμενη σε αίτημα των αρχών του Μαλή. Είδαμε ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σαχέλ ε, δεν έχει εφαρμοστεί σε όλες τις, τις διαστάσεις, έχει παραμείνει κυρίως σε επίπεδο ε, θεωρητικό, εγγράφων, επί χάρτου. Έχουμε πάρα πολλά έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλους τους τομείς και ενδεχομένως πολύ λιγότερες πράξεις τελικά επιτόπου. Νομίζω ότι ο κίνδυνος, ο υπαρκτός κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Αν η στρατιωτική επιχείρηση στο Μαλί είναι μικρότερη από αυτήν στη Λιβύη, τελικά ε, θα χάσουμε άλλη μια ευκαιρία να αντλήσουμε τα σωστά διδάγματα και θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την κατάσταση προκειμένου να εξάγουμε τα σωστά ε, συμπεράσματα ε, για το τι συμβαίνει. Και το λέω αυτό όχι μόνο γιατί το Μαλί ε, είναι μέρος μιας ευρύτερης περιοχής. Είδατε ότι την επίθεση στα σύνορα εντός Αλγερίας και συνορεύει και με τη Λιβύη. Όλα αυτά δημιουργούν μια πολύ ευρύτερη περιοχή την οποία θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως, αλλά θα πρέπει να δούμε και τις ευθύνες μας έναντι των Αφρικανικών κρατών γενικότερα. Ε, δεν ε, ενδιαφέρθηκαν να εμπλακούν άλλες διεθνείς δυνάμεις, ευρωπαϊκές δυνάμεις μεταξύ άλλων σε αυτή την ε, επιχείρηση, αλλά δεν έχουν και οι άλλοι εκτός Ευρώπης ε, το ίδιο ενδιαφέρον ε, με εμάς για αυτή την περιοχή. Νομίζω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Όλο και περισσότερες προκλήσεις θα υψώνονται μπροστά μας και θα είναι ευθύνη της Ευρώπης να ανταποκρίνεται και να στέκεται στο ύψος αυτών των προκλήσεων. Γι' αυτό είναι και εξαιρετικά σημαντικό να αντλήσουμε τα σωστά διδάγματα από την επιχείρηση στο Μαλή Να, κατά τα λοιπά, να δώσω το λόγο στον Συμπρόεδρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Γιώχαν. Δεν έχω και εγώ να πω πολλά πράγματα με τη σειρά μου. Νομίζω ότι όλοι παρακολουθήσαμε τις πρόσφατες εξελίξεις στο Μαλί. Να ευχαριστήσω τον στρατηγό ε, Ρουμπί, ο οποίος είναι σήμερα ε, μαζί μας. Δεν είναι ποτέ εύκολο για έναν στρατιωτικό που εκπροσωπεί συγκεκριμένη χώρα ε, μέλος να ε, έρχεται και να μας απευθύνει το λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί σίγουρα δεσμεύεστε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένη ε, ορολογία και γλώσσα αν θέλετε στην τοποθέτησή σας. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως το είδαμε και την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο, εμείς έχουμε κατανόηση και όχι μόνο κατανόηση, ε, αλλά στηρίζουμε εν γέννη τη δράση ε, της Γαλλίας στο Μαλί. Μπορεί να υπάρχουν ε, διαφορετικές φωνές, αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε στήριξη να παρουσιάσουμε και πιστεύουμε ότι αυτή η δράση αντικατοπτρίζει ε, την έλλειψη μιας συλλογικής ευρωπαϊκής δράσης, κάτι το οποίο θα είχαμε δικαίωμα, αν θέλετε, να ελπίζουμε από τη στιγμή που το Μαλί ε, είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό ε, παρόν στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σαχέλ, για την υποσαχάρη Αφρική γενικότερα. Μας εκπλήσει το γεγονός ότι εξεπλάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ισλαμιστική ε, επίθεση. Σε κάθε περίπτωση η Γαλλία είναι σαφές ότι ε, αντέδρασε εγκαίρως, γρήγορα, αλλά ε, θα μάθουμε περισσότερα γι' αυτό μετά την δική σας παρέμβαση. Πάρα πολλά ερωτήματα προκύπτουν για τη συνέχεια. Αυτό το οποίο περιμένουμε από εσά απόψε είναι να μας ενημερώσετε, να μας κάνετε ένα briefing για τις ε, επιχειρήσεις που βρίσκονται εν εξελίξη, για το βαθμό στον οποίο η Γαλλία είναι ικανοποιημένη με την επίτευξη των στόχων που είχε θέσει, ε, κάποιες πληροφορίες για τη διάρθρωση με, τις, με τα αφρικανικά στρατεύματα, γιατί αυτό έχει ζητηθεί και από τα ψηφίσματα τα δύο τα σχετικά του ΟΗΕ, ε, πώς υπάρχει η σύνδεση και διάρθρωση με την αποστολή εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το EUTM, Training Mission δηλαδή, πώς ε, ε, θα επιταχυνθεί ε, η εφαρμογή αυτής της αποστολής εκπαίδευσης ώστε να είναι πλήρως λειτουργική αλλά και όταν αυτό γίνει να μην θεωρηθεί ότι είναι το ενδεικτικό, το απολυτήριο που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποχωρήσει πλήρως από την περιοχή. Δεν είναι αρκετό δηλαδή το EUTM για να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει κάνει τη δουλειά της. Ε, να μας ε, ε, παρουσιάσετε και τις συνεισφορές των κρατών μελών ενδεχομένως, γιατί βλέπουμε ότι οι δυνατότητες, το δυναμικό αλλάζει και διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. υπάρχουν πολλές διαφορές και αυτό ενδεχομένως είναι ε, τροχοπέδι για την ε, θέσπιση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Περιμένουμε πολλά από εσάς, ε, είναι βέβαιο αυτό, στρατηγέ. Όμως Είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρετε. Ε, Βεβαίω δεν θα σας ζητήσουμε να μας αποκαλύψετε πληροφορίες που θεωρούνται απόρριτε και εμπιστευτικέ, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να μας διαφεωτήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη τιμή για μένα να παρεμβαίνω εδώ, να σας ε, απευθύνω το λόγο. Ε, παίρνω το λόγο ως ε, στρατιωτικός εκπρόσωπος της Γαλλίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Σίγουρα θα γνωρίζετε όμως ότι παρόλο που ανήκω και στις δύο και εκπροσωπώ τη Γαλλία και στις δύο οργανώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που έχω πραγματικά στην καρδιά μου συγκριτικά με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία βεβαίως. Ε, συνεργαζόμαστε στενά με τις ένοπλες ε, δυνάμεις ε, του Μαλή αλλά και με τις δυνάμεις της Αφρικανικής Ένωσης, τις Αφρικανικές δυνάμεις οι οποίες ήδη έχουν φτάσει επί τόπου. Και όλα αυτά εντάσσονται στο διεθνές ε, σκέλος των δράσεων και της Αφρικανικής Ένωσης και του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το περίπλοκο πλαίσιο λοιπόν στόχος μας ήταν με την παρέμβασή μας να αντιμετωπίσουμε επί κατεπηγόντως μία κατάσταση πρωτοφανή παρόλο που ήταν και προβλέψιμη αν θέλετε. Έχω διαβάσει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σαχέλ και στη δεύτερη τρίτη σελίδα βρίσκεται ένας χάρτης ο οποίος όταν ε, καταρτίστηκε το έγγραφο της στρατηγικής δείχνει ακριβώς την τοποθεσία, την ίδια τοποθεσία όπου σήμερα υπάρχει το πρόβλημα και όπου σήμερα τελικά ε, επεμβήκαμε μετά την, το ρητό αίτημα των αρχών του Μαλή και μετά την έγκριση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, η Γαλλία λοιπόν παρενέβη στρατιωτικά ε, στην χώρα αυτή και στις 11 Ιανουαρίου αποφάσισε να εμπλέξει τις γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση στο Μαλή θα ήθελα να σας δείξω ένα χάρτη και να τον έχουμε πάντοτε ε, σε προβολή ε, για να τον βλέπουμε γιατί νομίζω ότι είναι ε, καλύτερο για την ενημέρωση όλων μας. Θα ήθελα να σας μιλήσω λοιπόν για τις γεωστρατηγικές συνθήκες αυτής της παρέμβασης. 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η έκταση στο Μαλί, δύο φορές η Γαλλία. Το πιο στενό σημείο, ε, το βλέπετε στο χάρτη, είναι εκεί όπου μαχόμαστε αυτή τη στιγμή. Η, έκταση είναι η ίδια απόσταση όσο είναι από τον Μπογντό μέχρι το Στρασβούργο, 900 χιλιόμετρα από το βορρά στο νότο, 1800 χιλιόμετρα από την Ανατολή ω τη Δύση. Πρωτεύουσα είναι το Μπαμάκο, 4.500 χιλιόμετρα μακριά από τις Βρυξέλλες. Το, Μαλί είναι μια ε, χώρα περιτριγισμένη από άλλες χώρες, δεν έχει έξοδο, διέξοδο προς τη θάλασσα, έχει κοινά σύνορα με 7 χώρες τις οποίες ε, βλέπετε ε, στο χάρτη και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μια πολύ σημαντική από στρατιωτικής πλευράς λεπτομέρεια. Το γεγονός ότι ε, το κλίμα χαρακτηρίζεται από τις περιόδους ξηρασίας και ε, τις υγρές περιόδους υγρασίας. Υπάρχουν εποχές όπου δεν μπορούμε καμία στρατιωτική δράση να αναλάβουμε. Σε καμία περίπτωση. Για να στείλουμε μια δύναμη στα 4.500 ε, χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες σε μια τόσα ευρεία έκταση γεωγραφική ε, τελικά πρέπει να αποστείλουμε εκατοντάδες τόνους υλικού, καυσίμων, ε, ε, εφοδίων πάρα πολλά αεροσκάφη, πάρα πολλέ πτήσει ανεφοδιασμού δηλαδή ε, σε πολλαπλά επίπεδα. Απέναντί μας έχουμε τρομοκρατικές ομάδες αποφασισμένες, συνηθισμένες να δρουν σε τέτοιες τόσο δύσκολες περιοχές ε, και πολύ καλά εκπαιδευμένε. Έχουμε καταρχά το ΑΚΙΜ, την Αλκαΐδα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ, έχουμε το ε, κίνημα για την ενότητα και το τζιχάτ στη Δυτική Αφρική και έχουμε και το Ανσαντίν, ε, τους υπερασπιστές του Ισλάμ. Αυτά είναι ε, τα τρία σκέλη, αν θέλετε, τις, οι τρεις ομάδες οι τρομοκρατικές ε, που δρούν και γνωρίζαμε άλλωστε ότι ήταν ενεργές εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ονομάσαμε την ε, γαλλική στρατιωτική επιχείρηση σε πάλι, είναι μια μικρή αλεπού της ερήμου αυτή και ε, ο στόχος είναι τριπλός. Πρώτον, να σταματήσει η επίθεση των ε, τρομοκρατικών ομάδων οι οποίες κατέβαιναν από το βορρά προς τα, προς δυτικά και προς τα ανατολικά με τελική κατεύθυνση των παμάκο να συμβάλλουμε στη διατήρηση της εδαφικής συνέχειας του Μαλή, να επιτρέψουμε την λήψη διεθνών αποφάσεων ως προς την ανάπτυξη της αφρικανικής δύναμης και ως προς την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αποστολής Εκπαίδευσης στο Μαλί, το, του EUTM δηλαδή. Οι εθνικές μας ένοπλες δυνάμεις ε, ε, έχουν τέσσερες αποστολές. Πρώτον, να βοηθήσουν τις ένοπλες δυνάμεις του Μαλή να σταματήσουν την έλευση των τρομοκρατών με αεροπορικές επιδρομές αλλά και με χερσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, να ε, βομβαρδίσουμε ε, τις ε, βάσεις των τρομοκρατών για να τους εμποδίσουμε να κάνουν νέες επιθέσεις. Τρίον, τον, να επιτεχύνουμε την, την ανάπτυξη των αφρικανικών ε, δυνάμεων του αμίσμα και τέλος, δηλαδή της στρατιωτικής αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στην Σομαλία, και τελικά μαζί με τη, τις ένοπλες του Μαλή σταματήσαμε την έλευση των τρομοκρατών, την κάθοδό τους προς τον Μπαμάκο. Βλέπετε ε, το πιο στενό κομμάτι του Μαλή στο χάρτη και εκεί στην Τουέντζα ήταν ε, το μέρος όπου δράσαμε. Δυτικά ε, έχουμε τον Διαμπαλή και το Εναρά νότια στη δεξιά γωνία της Μαυριτανίας, τα σύνορα με το Μαλί, εκείνη η περιοχή όπου δρούμε κυρίως. Ποια είναι τώρα η ανθρωπιστική κατάσταση. Ε, ε, επιδεινώνεται διαρκώς. Έχουμε μετακινήσεις αμάχου πληθυσμού που προσπαθεί να φύγει από τις επικίνδυνες περιοχές, μαζικές ε, εξόδους προς τον Ήγυρα, την Μπουρκίνα Φάσο, τη Μαυριτανία και την Ιγυρία από πλευράς αμάχου πληθυσμού. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, το UNHCR, την ύπατη αρμοστία για τα για τους πρόσφυγες. Έχουμε σήμερα 2.000 ε, ε, πρόσφυγες 50.000 στον Ήγυρα, 38.000 ε, στην Πουρκίνα Φάσο, πολλές χιλιάδες δηλαδή στις γειτονικές χώρες γενικά. Ως προς τις τρομοκρατικές ομάδες, ε, πρέπει να σας πω ότι προσπαθήσαμε να εμπλέξουμε τις ένοπλες δυνάμεις του Μαλή όσο το δυνατόν περισσότερο και έτσι οι τρομοκρατικές ομάδες υποχώρησαν, ε, υποχώρησαν σε σχέση με τη ζώνη επαφής που είναι στα στενά που βλέπετε στο χάρτη και κυρίως στην πόλη του Τιμπουκτού, στην πόλη του Γκάο. Ε, δεν ξέρω αν τη βλέπετε στο χάρτη και στην πόλη του Κιντάλ, η οποία είναι πολύ βόρεια κοντά στην Αλγερία αλλά και σε ένα ε, τέταρτο ε, σημείο αρκετά κοντά στα σύνορα με τη Μαυριτανία πάντοτε στο βορρά. Οι αφρικανικές δυνάμεις όλο και περισσότερο πληθαίνουν ε, δεν ξέρω αν θέλετε να σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες για το δυναμικό που έχουν αναπτύξει επί τόπου. Έχω στοιχεία, μπορώ να σας τα δώσω εάν μου θέσετε τις αντίστοιχες ερωτήσεις στη συνέχεια. Δέκα αφρικανικές χώρες στελεχώνουν αυτές τις αφρικανικές ένοπλες δυνάμεις που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Είναι σε φάση ανάπτυξης λοιπόν στο Μπαμάκο. Έχουν επιταχυμένο χρονοδιάγραμμα συγκριτικά με αυτό που είχαν προγραμματίσει εξ αρχής. Και ε, σε τέλος, θα πρέπει μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις του Μαλή να επανακατακτήσουν το βορρά της χώρας αυτής ώστε να εδρεωθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις και να ξεκινήσει η κατάλληλη πολιτική διαδικασία για την διεξαγωγή εκλογών στη χώρα αυτή ώστε να εκλεγεί νόμιμη κυβέρνηση. Πάντοτε ε, με πλήρη σεβασμό ε, στα ε, ψηφίσματα του ΟΗΕ και το τελευταίο το οποίο είναι το 2085. Επομένως, η Νιγηρία, η Σενεγάλη, το, το Γκό και η Μπουρκίνα Φάσο ε, ε, είναι οι χώρες όπου έστειλαν τις πρώτες στρατιωτικές δυνάμεις στο Μαλί και προβλέπεται ε, να στείλουν δυνάμεις ένοπλες και ο Νίγηρας, η Γουινέα, η ακτή του Ελεφαντοστού, το Τσάντ και το Μπενίν. Ως προς τον εξοπλισμό τους, είναι δύσκολο το θέμα αυτό και η δυνατό, προσπαθούμε να τους διευκολύνουμε όσο να το περισσότερο ε, θέλουμε οι αφρικανικές δυνάμεις να είναι ώστε να τον νωρίτερα και όσο να τον πιο γρήγορα ε, λειτουργικές και επιχειρησιακές. Στις 29 Ιανουαρίου στην Αντίς Αμπέμπα θα λάβει χώρα μια διάσκεψη των δωρητών ώστε να υπάρξουν κονδύλια και να συγκεντρωθούν κονδύλια για να εξοπλιστούν καλύτερα οι αφρικανικές ανοπλές δυνάμεις. Και ελπίζουμε ότι με αυτή την ευκαιρία της διάσκεψης των δωρητών θα ε, υπάρξει εκεί μια δεύτερη ε, συνεδρίαση ε, υπέρ του εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων του Μαλή. Περιμένοντας λοιπόν να είναι πλήρως επιχειρησιακές οι αφρικανικές δυνάμεις, ένοπλες δυνάμεις, οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις εν τω μεταξύ έχουν την εντολή να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν την κατάσταση έτσι όπως είχε πριν από τις Ισλαμιστικές επιθέσεις και να παραμείνουν όσο χρειάζεται και όσο χρειαστεί ώστε να αποκατασταθεί με βιώσιμο τρόπο η πρώτερη κατάσταση ε, στο Μαλί, έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να ληφθούν ε, διεθνείς αποφάσεις, δηλαδή να αναπτυχθεί η αφρικανική δύναμη και να αναπτυχθεί και η ε, αποστολή εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαλί, όπως σας είπε προηγουμένως και ο στρατηγός Ντεγούσιε. Ο στρατηγός Λεκουάντ, ο οποίος είναι επικεφαλής του EUTM, ήταν σε αναγνωριστική αποστολή και γι' αυτό δεν είναι σήμερα μαζί μας, για να αναγνωρίσει ποιες είναι οι ανάγκες εκπαίδευσης. Θα επιστρέψει σήμερα το βράδυ και θα μας βοηθήσει να ε, αξιολογήσουμε ε, ποια είναι αυτά τα οποία ε, χρειάζονται. Σε αυτό το στάδιο δεν έχω προβλέψει να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά με χαρά θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Το προνόμιο του Προέδρου να ρωτήσω πρώτος. Μια ερώτηση επί των ε, γεγονότων. Έχετε μια συγκεκριμένη αξιολόγηση του μηχανισμού και των εξοπλισμού που διαθέτουν οι Ισλαμιστικές ε, ενόπλες ε, δυνάμεις ε, έχει γίνει κάποια αξιολόγηση σοβαρή σχετικά με αυτές τις τρομοκρατικές ε, ομάδες. Φαίνεται ότι ε, αυτά που διαθέτουν είναι πέρα από αυτά που είχαμε σκεφτεί και ότι ο εξοπλισμός τους είναι πολύ πιο ε, εξυζετημένος από ό,τι θεωρούσαμε. Και μια πιο πολιτική ερώτηση. Το βασικό ερωτηματικό είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, όλοι είχαν προβλέψει μια στρατιωτική επιχείρηση για να μπορέσουν να επαναφέρουν την ακεριότητα στο δεύτερο μέρος ε, του 2013, όχι πριν. Όμως ε, λόγω της επίθεσης των Ισλαμιστών ε, άλλαξαν τα πράγματα. Πήγαν πιο γρήγορα. Πώς ε, θα μπορέσουμε αυτή την καθυστέρηση των έξι μηνών σε επιχειρησιακό στάδιο να την αναπληρώσουμε. Γιατί είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα και πραγματικά είναι σημαντικό γιατί ε, καθορίζει και την ακολουθία των γεγονότων. Η κάθε ομάδα έχει το λόγο. Ο Ιλιαν Πάσκου είναι ο συμπρόεδρος και είναι ο πρώτος που θα κάνει ερώτηση. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι κάθε τέτοια επιχείρηση όταν ξεκινάει, έχει τουλάχιστον σχεδιάσει σε γενικές γραμμές τον... την έξοδο διαφυγής. Πώς θα τελειώσει το όλο πράγμα. Εδώ υπάρχουν ε, στρατιωτικά και πολιτικά καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν. Ο νέος στρατός του Μαλή θα πρέπει να είναι στρατιωτικά αποτελεσματικός και πολιτικά ελεγμένος, γιατί ιδάλλως ε, θα έχουμε ένα κανόνι που θα είναι έτοιμο να πυρσοκροτήσει να στη στιγμή και να φέρει ε, τους πάντες στο σημείο μηδέν ευθύς εξ αρχής. Δεύτερον, η πολιτική διαδικασία ίσως να μην είναι επαρκής ε, για να παγιωθεί η εντολή των θεσμών. Ίσως πρέπει να υπάρχει κάποια παρουσία λοιπόν που να χρειάζεται. Χρειάζεται παρακολούθηση όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο, γιατί φυσικά αυτό το έδαφος είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί, αλλά και πολιτική αποπτία και παρακολούθηση χρειαζόμαστε. Πολιτική επιτήρηση μάλλον το στοιχείο το βασικό που πρέπει να σκεφτούμε για το τέλος της επιχείρησης είναι η υπεράσπιση των στρατηγικών στόχων. Δεν ξέρω αν η αποστολή εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ξεπεράσει το καθήκον της εκπαίδευσης ε, του ε, στρατού του Μαλή, να δημιουργήσει ένα πυρήνα, ας πούμε, που θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ή θεωρείτε ότι πρέπει να μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναλάβει τα υπόλοιπα καθήκοντα. Αυτά στα οποία δηλαδή θα συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για τις διάφορες ε, πολιτικές ομάδες τώρα οι εκπρόσωποι θα μιλήσουν. Ο κύριος Γκάλερ για το ΕΛΚ. Ναι, ευχαριστώ. Παρακαλώ, προσοχή γερμανικά. Καταρχάς να σας ευχαριστώ. Είστε ο εκπρόσωπος της Γαλλίας και θεωρώ ότι η Γαλλία ε, προς το συμφέρον όλων με ή χωρίς εντολή ανέλαβε την ευθύνη. Ελπίζω ε, να αλλάξει και η στάση της κυβέρνησής μου τις επόμενες ημέρες, δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη και υποστήριξη και γενικά μια υποστήριξη όχι μόνο γλωσσική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μια πιο γενική υποστήριξη και ελπίζω πολλά τα κράτη-μέλη όταν έχουν τη δυνατότητα να μην αφήσουν μόνο τη στην Γαλλία. Η πρώτη ερώτηση. Πόσο μπορείτε να εκτιμήσετε ότι από μόνοι σας θα μπορέσετε να αντέξετε είναι μια περιοχή δυόμιση φορέ μεγαλύτερη από τη Γαλλία. Πρέπει να καλύψετε τεράστιε εκτάσει. Ε, πόσο μπορείτε να το κάνετε αυτό. Μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό ε, θα ασκούσε ίσως πίεση και στα άλλα κρατημέλη. Άλλη μια ερώτηση που ε, ακολουθεί τον Συνάλφο Πάσκο. Στον στρατό του Μαλή και στην κυβέρνηση ε, ποιοι είναι αυτοί που συνομιλείτε, είναι αυτοί που κάνανε το ε, πραξικόπημα, γιατί η κατάσταση είναι λίγο περίεργη. Είναι ένας ε, νόμιμος στρατιωτικός εταίρος αυτός που συνομιλείτε; Τρίτη ερώτηση. Ήδη υπάρχει κάποια εμπειρία σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται ο λαός στο Μαλί την γαλλική παρουσία. Είναι θετική δηλαδή η διάσταση, η διάθεση και από τους εχμαλώτους. Πώς είναι η χρηματοδότηση σε αυτούς τους ε, αντάρτες, από πού προέρχονται τα χρήματα, πώς είναι η αλυσίδα πληρωμών. Είναι έξω από το μαλλί. Ε, υπάρχει πρόσβαση σε μέσα άμεσα εκτός μαλλί. Πώς θα μπορούσαμε να τους αποκόψουμε από αυτούς και στρατιωτικά και οικονομικά. Ευχαριστούμε για τους ε, σοσιαλδημοκράτες η κυρία Κόπα. Κοπά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον στρατηγό. Θα ακολουθήσω τον συνάδελφο Πασκού σχετικά με τα εξή θέματα. Η μεγάλη πρόκληση είναι να βρούμε μια ε, βιώσιμη και ειρηνική λύση στο Μαλί. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, είναι τεράστιο το έδαφος, είναι τεράστια και η πρόκληση. Η Γαλλία δήλωσε ότι δεν έχει την πρόθεση να παραμείνει στο Μαλί μετά το τέλος των εχθροπραξιών. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το Μαλί δεν θα γίνει κέντρο των τρομοκρατών. Η επόμενη μέρα πραγματικά θα είναι η μεγάλη πρόκληση. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα τελειώσουν κάποια στιγμή και μετά τι θα γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι το Μαλί δεν είναι μόνο γαλλική υπόθεση, είναι ε, υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω κάποιες συγκεκριμένες ε, ε, ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση στα βόρεια του Μαλί, γιατί εκεί γνωρίζουμε ότι συνεχώς υπάρχουν ε, προβλήματα με τους Τουαρέγκ. Ε, υπήρχαν εξεργέσεις, η τελευταία ήταν το 2006 και είναι ένα θέμα που εντάθηκε μετά την πτώση του καθεστώτος Καντάφη. Μπορεί να είναι και σχεδιασμένη γιατί όλοι γνωρίζουν ότι ο στρατός της ε, Λιβύης έχει εκπαιδευτεί από άτομα που ε, δημιουργήθηκε μάλλον από άτομα που ήταν στο Σαχέλ και μετά από την πτώση του Καντάφη έχουν ένα ρόλο όπως έγινε και με τον στρατό του Σαντάμ Χουσέιν που ξεκίνησαν τρομοκρατικές δράσεις μετά την πτώση του. Τώρα για τα ε, στρατιωτικά εργαλεία. Ε, τι έχουν στα χέρια τους οι αντάρτες και οι τρομοκράτες, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να έρθουν ε, και εδώ γιατί δεν έχει ελεγχθεί η Λιβύη σε επίπεδο στρατιωτικό ακόμη. Δεύτερη ερώτηση σχετίζεται με την υποστήριξη που προέρχεται από την Αφρικανική Ένωση και συγκεκριμένα από χώρες όπως η Σενεγάλη για παράδειγμα, η οποία είναι πολύ καλά εξοπλισμένη για να γίνει βάση υποστήριξης για το Μαλί. Και συνήθως υπάρχει παράδοση με ε, τη Σενεγάλη και τη Μαυριτανία σε επίπεδο συνεργασίας χρήσιμης για τη Γαλλία. Ευχαριστούμε η κυρία Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ στρατηγέ που είστε μαζί μας, ε, που, θα μας, που μας εκθέσατε τα πολύπλοκα αυτά ε, δεδομένα. Οι συνάλφοι έκαναν αιχμηρές ε, ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον, το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο. Εγώ Επίσης έχω και κάποιες ερωτήσεις για το πρόσφατο παρελθόν και άμεσο μέλλον. Να πω ότι στην τελευταία ολομέλεια στο Στρασβούργο εξέφρασα εκ μέρους της ομάδας μου και της χώρας μου, του Βελγίου, την υποστήριξή μας, την αρχική υποστήριξή μας στην πρωτοβουλία της Γαλλίας που ε, πήρε τα Ινία. Ε, στο ενδιάμεσο διάστημα ξεχνάμε ότι εδώ και μήνες ε, η κυβέρνηση και οι διάδοχοι τους στο Μαλή αρνούνταν οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση. Έτσι λέγανε τουλάχιστον. Και πραγματικά δεν πώς μπορούσαμε να πιστέψουμε τότε ότι θα πάμε σε άλλο επίπεδο. Σήμερα εντάξει, μπορεί να λέμε ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία, καλά είναι να ξεκινήσουμε να δρούμε, αλλά τι μπορεί αυτό να σημαίνει στο μέλλον σε παρόμοιες καταστάσεις. Επιπλέον υπάρχει ένα άλλο θέμα που αναρωτιέμαι. Τι συμβαίνει, ίσως ε, όμως δεν θα αντιθέσω γιατί την απάντησε ο προηγούμενος ε, ο μιλητής, ε, και θα τη θέσω και σε εσά. Η εκοφαντική σιωπή του ΝΑΤΟ. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Διαβάζω σε κάποιες ε, εφημερίδες επίσης ότι οι Αμερικανοί για μια μεγάλη χρονική περίοδο αναγκάστηκαν να εκπαιδεύσουν τις δυνάμεις ε, του Μαλή, να τις ε, εξυγχρονίσουν και αυτό τους κόστησε δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια και αυτές οι δυνάμεις πέρασαν στην άλλη πλευρά τελικά. Είναι αλήθεια αυτό. Και αν όντω, τι θα κάνουμε ή τι σκεφτόμαστε να κάνουμε για να αποφύγουμε μια επανάληψη αυτού του φαινομένου. Τέλος. Ακούω πολλές φορές και δεν αμφιβάλλω ότι κάποιοι δορυφόροι μπορούν να δουν που βρίσκονται ε, οι διάφορες ε, πολιτικές ε, τρομοκρατικές ομάδες. Αναρωτιέμαι, σκεφτόμαστε έναν προληπτικό ε, πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Ε, δηλαδή, ε, αν ξέρουμε κάπου ότι υπάρχει μια τρομοκρατική ομάδα, αν μπορούμε να πάμε και να την εξουδετερώσουμε. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Και τι θα γίνει με τον πολλαπλασιασμό τέτοιων ομάδων. Νομίζω ότι αυτά είναι ερωτήματα που πραγματικά πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν προετοιμάζουμε το μέλλον. Τέλος, ο πρόεδρος τη Γαλλική Προεδρίας είπε ότι η επιχείρηση θα διαρκέσει όσο θα χρειαστεί. Κατανοητό, αλλά είδαμε σε εσωτερικές ε, περιπτώσεις ε, πόσο μία ε, απελευθερωτική δράση τελικά γίνεται κατοχή. Αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Και τέλος η κυρία Λούνετσεκ. Όχι, κυρία Κέλμινσεν. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, στρατηγέ, για την παρουσία σας εδώ. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα ειδική στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και γι' αυτό δεν θα μπω σε αυτά τα χωράφια. Ακόμα και αν ακολουθώ, παρακολουθώ την ε, επικαιρότητα, ξέρω το μαλή, ξέρω την περιοχή, την παρακολουθώ σε κάθε χωριό τι συμβαίνει. Αυτό που με ανησυχεί στην ε, Υποεπιτροπή επίση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπου συμμετέχω, είναι οι άντρε και οι γυναίκες που ζουν στα βόρεια του Μαλή. Ε, καταρχάς ε, υπάρχει πρόσφατη δήλωση της Αφρικανική Αφρικανικής Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μιλά για την αύξηση του εκτοπισμού πληθυσμού τις τελευταίες ημέρες και ζητά η Επιτροπή αυτή να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για να μπορέσουν να κινηθούν εσωτερικά οι εκτοπισμένοι. Δηλαδή ο στρατός να εμπλακεί για να επιτρέψει στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να είναι ασφαλείς και να διασφαλίσουν αυτούς τους διαδρόμους. Δεύτερον, πάλι οι μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις όπως το Human Rights Watch ε, αναφέρουν ότι υπάρχουν εθνικές, ε, εθνικιστικές εντάσεις που έχουν επιδεινωθεί στα βόρεια του Μαλή. Υπάρχουν φόβοι, όπως για παράδειγμα στο Τιμπουκτού ο, ο Δήμαρχος είπε ότι ανησυχεί για αντίπεινα. Μετά από την άφηξη στο βορρά των Αφρικανικών στρατευμάτων, είπε. Τέλο πάντων, εγώ θεωρώ ότι πρώτο φόβος ήταν ο γαλλικός στρατός, αλλά τέλος πάντων εθνικιστικές εντάσεις. Εγώ θέλω να μάθω ποιο είναι ο ρόλος που θέλετε να παίξετε. Ίσως ενδιάμεσες δυνάμεις θα ήταν ιδανικό, αλλά ας μην το μιλάμε αυτό. Είναι ε, μια κατάσταση που τη γνωρίζω καλή, στο Μαλί, όπως μου λένε. Αυτή τη στιγμή έχουν μίσος ε, εναντί του MNLA που συμμετείχε τον ε, Ιανουάριο του 2012 στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, στις εχθρότητες κτλ. Να μην ξεχνάμε όμως ότι είναι και μια πολιτική οργάνωση ταυτόχρονα. Και ο εισαγγελέας του Διεθνούς Δικαστηρίου ε, ξεκίνησε μια έρευνα από το 2012 για όλες αυτές τις οργανώσεις, ε, για το στρατό, ε, για τις παραστρατιωτικές οργανώσεις που υπάρχουν εκεί. Όλα αυτά είναι ανησυχητικά. Όλα αυτά λοιπόν με ανησυχούν. Δεν πρέπει να συγχαίουμε ε, τους ανοιχτόχρωμους και τους σκουρόχρωμους ε, και, μια άλλη, ε, και όλες αυτές τις οργανώσεις. Ε, στο βορρά υπάρχει ακόμα ρατσισμός, υπάρχουν μαύροι σκλάβοι και πραγματικά υπάρχουν πολλοί φόβοι. Ποιο είναι ο ρόλος που θα μπορούσε να παίξει ο γαλλικός στρατός για να αποφύγουμε στα βόρεια του Μαλή να υπάρχουν αντίπεινα και ακραίες αντιδράσεις. Ευχαριστούμε. Τέλος ο Τσάρλ Τάνοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω κύριε στρατηγέ. Η ομάδα μου, η ΣΥΑΡ, ε, που έχει ένα μεγάλο βρετανικό συντηρητικό κομμάτι. Χαίρεται για την γαλλική συμμετοχή στο Μαλί και χαιρόμαστε που ο Κάμερον έχει προτείνει μια ε, συμμετοχή της Βρετανίας ε, Ήθελα να σας ρωτήσω μια σειρά πράγματα. Πρώτον, ένα από τα πράγματα που με ανησυχεί και φυσικά είναι και εθνικό γαλλικό συμφέρον, είναι ε, τα ορυχεία κοντά στον Ήγηρα. Ουράνιο. Έχουν ουράνιο. Αν η τζιχάντ πάρει τον έλεγχο εκεί ειδικά ε, του ουρανίου που θα μπορέσει να δημιουργήσει μια ε, ατομική βόμβα που θα μπορούσε να απειλήσει στις ε, πόλεις της Ευρώπης γιατί είμαστε τόσο αργοί στην κινητοποίηση των αφρικανικών στρατευμάτων. Είχαμε στις 13 Δεκεμβρίου κάποιες λίγες μονάδες και μετά ξαφνικά λόγω της πήγουσας κατάστασης είχαμε τόση πολλή συμμετοχή. Επίσης, το ΝΑΤΟ με αυτή την ε, ε, ασπίδα τη βορειοατλαντική και που θα μπορούσε να καλύψει και το κέρας της Αφρικής. Είναι αλήθεια ότι το ΝΑΤΟ δεν θέλει να συμμετάσχει. Πήγε στη Λιβύη αλλά δεν θέλει να πάει παραπέρα. Πέρα από αυτό δηλαδή που κάνει ε, στη Σομαλία αυτή τη στιγμή κατά της πειρατείας. Και επίσης το EUTM που τώρα θα ενισχυθεί και θα επιταχυνθεί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ε, στο Μαλί και σε άλλες αφρικανικές χώρες. Αυτά είναι μεγάλα θέματα που μας ανησυχούσαν και στην Ουγκάντα με την αποστολή ε, εκπαίδευσης. Υπήρχαν πολλές αυτομολύσεις στο Αλσαμπάμ και πώς δεν ξέρουμε ότι οι στρατιώτες του Μαλί δεν θα πάνε με τους Ισλαμιστές. Άκουσα ότι υπάρχουν κάποιοι στο Ακίμα και στο Αλσαντίμα που ε, προέρχονται από το στρατό του Μαλί και μπορείτε να μας δώσετε και κάποια ιδέα για το μέγεθος του εχθρού σας. Δηλαδή, πόσοι ένοπλοι μαχητές ανήκουν σε αυτές τις τρεις ε, ε, οργανώσεις και τις πιο εξτρεμιστικές που αναφέρθηκαν. Μιλάμε για νούμερα από μερικές εκατοντάδες μέχρι και μερικές χιλιάδες στο ίντερνετ. Και υπάρχουν κάποιοι που δρούν και στην Αλγερία. Και τέλος, αυτό που είπε και η πράσινη συνάδελφος, στο MNLA, ε, συζητήσαμε γι' αυτό πριν από ε, λίγο καιρό, που στην αρχή ήταν πολιτική οργάνωση, μετά έγινε ένοπλη. Είναι ουδέτερη ή είναι με τους ε, ε Ισλαμιστές και είναι εναντίον των Γάλλων. Μπορούμε να τους εκλογικεύσουμε, να μην ε, μάχονται και μετά να βρούμε μια πολιτική λύση και τελικά να έχουμε και μια συνένεση για κάποια αυτονομία στο Βορρά και στην ε, μειοψηφία του του ΑΡΕΓ. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση, η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε σε αυτή την Επιτροπή και πάλι εκ μέρους της ομάδας μας των Πρασίνων Πολύ καλωσορίσαμε τα βήματα που έκανε η γαλλική κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, πολύ εξημών αναφερθήκαμε και στα προβλήματα τα οποία δεν είχαν εξεταστεί στο παρελθόν. Όχι από το γαλλικό στρατό φυσικά, αλλά από εμάς ως Ευρωπαίους, ε, από εμάς ως Ευρωπαίοι πολιτικοί. Το Μαλί ήταν ε, μια δημοκρατική χώρα και είχε και εκλογές για πολλά χρόνια, αλλά ποτέ δεν σκεφτήκαμε ε, τα θέματα του νεποτισμού της διαφθοράς ε, που υπήρχαν στη χώρα. Και πραγματικά δεν ξέραμε πώς θα προχωρήσει η κυβέρνηση και θα αντιμετωπίσει την ανέχεια που υπάρχει και το χάσμα μεταξύ των δύο μερών της χώρας που φαίνεται ότι υπήρχε πάντοτε. Υπάρχουν κάποια θέματα που σχετίζονται με τις μάχες που γίνονται και με αυτά που ήδη <laughs> ανέφερε η συνάδελφος. Το φόβο ότι μπορεί να υπάρχουν αντίπεινα καθώς προχωρούν οι δυνάμεις προς το βορρά. Επίσης υπάρχουν και κάποιες άλλες ανησυχίες ότι κάποια στοιχεία του στρατού του Μαλή και κάποιοι παραστρατιωτικοί που ήταν πιστοί ε, στον Τσιπρίν Τριάλο, Μπραχήμ Τριάλο και στο στρατό του Μαλή, που ήδη έχουν ε, διαπράξει εγκλήματα πολέμου κατά των ε, αμάχων στην περιοχή. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι αυτά τα εγκλήματα δεν θα συνεχιστούν και μετά, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα να γίνονται τέτοια πράγματα. Δηλαδή, το μέλλον μετά την στρατιωτική παρέμβαση θα είναι ακόμα πιο δύσκολο αν ε, δεν λάβουμε υπόψη ότι μπορεί να υπάρχουν ε, εγκλήματα και από τις δύο πλευρές. Και επίσης, ε, έχω ακούσει ότι αυτή η αποστολή, το έχουμε έχει ε, πολύ καλά προετοιμαστεί έχει γίνει κοινή εκπαίδευση. Ε, τι ξέρετε γι' αυτό. Μια άλλη ερώτηση που αναφέρεται στο μέλλον. Τι θα γίνει όταν απελευθερωθεί το έδαφος, όταν δεν θα είναι εκεί οι Γάλλοι. Υπάρχει κάποιο σχέδιο. Και για να επανέλθω σε αυτό που είπα στην αρχή, ε, ήδη ε, συζητάτε με άλλους σε πολιτικό επίπεδο επιτόπου τι θα γίνει μετά την παρέμβαση. Το Μαλί έχει ιστορία και παράδοση μιας κουλτούρας διαλόγου και επίλυσης διαφορών μεταξύ των διαφορών εθνοτικών ομάδων. Είναι κάτι που συνέβη, υπάρχει μια καλή παράδοση εδώ και χρόνια. Ο φόβος μου και φόβος πολλών είναι ότι σε άλλες χώρες όπως το Αφγανιστάν, Λιβύη, Ιράκ, όπου έγιναν τέτοιες παρεμβάσεις, παρόλο που τις χαιρετήσαμε, το ότι κερδίσαμε τον πόλεμο δεν σήμαινε ότι κερδίσαμε και την ειρήνη μετά. Αν τα θεσμικά προβλήματα που είναι βαθιά ριζωμένα στο Μαλί δεν λυθούν με τους ε, ντόπιου, τότε πραγματικά μπορεί να κερδίσουμε τον πόλεμο και να χάσουμε την ειρήνη. Και αυτό ε, πρέπει να το εμποδίσουμε και είναι προς συμφέρον μας. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριο Παντζέρη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πω αμέσως ότι στήριξα και στηρίζω την παρέμβαση της Γαλλίας, την επέμβαση της Γαλλίας ε, στο Μάλι. Πιστεύω και ίσω να μην είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή, αλλά θα χρειαστεί να επανέλθουμε από πολιτική άποψη στην υπόθεση αυτή, γιατί θα αρκούσε να δώσουμε το παράδειγμα της μετακίνησης ε, του ράλι Παρίντα Κάρ εδώ και κάποια χρόνια για να πούμε ότι έχουμε κάνει ένα σωρό λάθη όσον αφορά την πολιτική ασφάλεια τη περιοχή αυτή. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να εμβαθύνουμε στα λάθη του παρελθόντος γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να μην αποκομίσουμε διδάγματα. Θέλω να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτη παρέμβαση. Η επέμβαση στη δυτική έχει στόχο να νικήσει ή να περιορίσει τους ε, επαναστάτες. Γιατί στην ουσία τι, θα, ε, τι σημαίνει αυτό, ότι αν θέλουμε να τους νικήσουμε θα, θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι τέλους. Ε, εν πάση περιπτώσει, αν η στρατική επέμβαση λειτουργήσει, ο, ο κίνδυνος είναι να υπάρξει διάχυση αυτών των επαναστατών σε γειτονικέ χώρες, όπως ας πούμε για την Αλγερία. Έχει στρατό στα σύνορα ή στον Ήγηρα ή στη Μαυριτανία. Έχετε επαφές με αυτές τις χώρες ώστε να μπορέσετε να εμποδίσετε κάτι τέτοιο. Δεύτερη παρατήρηση για τον Ήγηρα. Πολλοί έγραψαν ότι είναι μια χώρα κάπως αμφίβολη γιατί από αυτή τη χώρα έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια τεράστια οπλοστάσια που προέρχονται από τη Λιβύη και συνεχίζεται αυτό το στρατιωτικό αυτή η στρατιωτική παρέλαση. Υπάρχει έλεγχος και ο Νίγηρας ανταποκρίνεται θετικά. Τέλος για το κίνημα απελευθέρωσης, το απελευθερωτικό κίνημα του Αζαγουάντα. Πολλά, πολύ, ε, εκπρόσωποι έγιναν δεκτοί και στο Παρίσι. Αν στην διαδικασία διαχωρισμού του μετόπου των, μάλλον διχασμού του μετόπου των επαναστατών ε, υπάρχει προσπάθεια για διχασμό και αυτό του ώστε να υπάρξει διαχωρισμός των τρομοκρατικών ομάδων από το απελευθερωτικό κίνημα. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο, στο ίδιο καλάθι και δεν θα πρέπει να δοθούν στοιχεία στους τρομοκράτες και να μην ε, ε, προεξοφλήσουμε ότι το ΆΡΕΓ είναι μαζί τους. Είναι, πρόκειται για στρατηγική, πολιτική και ε, στρατηγικής σημασίας. Σας ευχαριστώ πολλά ερωτήματα, <laughs> κύριε Υπουργέ, ε, κύριε Στρατηγέ, συγγνώμη. Ε, λίγο χρόνο έχετε να ε, απαντήσετε, αλλά θα πρέπει να μιλήσετε επί της ουσίας. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας και σας ευχαριστώ και για την υποστήριξη ε, που μας προσφέρεται και βλέπω ότι είναι γενικευμένη η στήριξη αυτή. Ξέρετε, ο Κλεμονσό στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είπε στον αρχηγό του επιτελείου του το εξής. Το ο πόλεμος είναι κάτι το εξαιρετικά σοβαρό για να το εμπιστευτούμε στους στρατιωτικούς και εμείς ίσως θα μπορούσαμε να, να το αντιστρέψουμε αυτό και να πούμε σήμερα ότι η ειρήνη είναι κάτι το εξαιρετικά σοβαρό για να το εμπιστευτούμε μόνο στους διπλωμάτες. Πάρα πολλές ερωτήσεις που θέσατε, θα προσπαθήσω να απαντήσω συνολικά σε όσο περισσότερο μπορώ. Να, να σας πω εξ αρχής ότι μου φαίνεται ότι έχετε υπερβολικές προσδοκίες, πολλές προσδοκίες από εμένα. Καλό νέο είναι αυτό. Και με τα μέσα όμως που έχουμε στη διάθεσή μας, με 2.500 ανθρώπους ε, και θα έχουμε 3.300 Αφρικανούς και 4.000 ή 5.000 ε, στρατιώτες από το Μαλί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε μια χώρα 14 εκατομμυρίων ε, κατοίκων. Άλλωστε ε, πάντοτε κανείς θα κάνει ό,τι μπορεί. Ε, Τούτων λεχθέντων, πολλές ερωτήσεις θέσατε. Ποιος είναι ο αντίπαλος που έχουμε συγκεκριμένα απέναντί μας. Να σας πω ότι έχουμε έναν αντίπαλο τον οποίο αξιολογούμε ε, βάζοντας τα κομμάτια του παζλ από τις εικόνες που έχουμε από το δορυφόρο, από τις εικόνες που έχουμε με τις χερσαίες δυνάμεις με τις οποίες έχουμε αγωνιστεί, τις οποίες έχουμε πολεμήσει επί τόπου. Δύο με τρεις χιλιάδες λοιπόν τρομοκράτες, τζιχαντιστές, δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, ποιο είναι ο πιο κατάλληλος όρος. Ε, στον άτομα μας αμφισβητούν την χρήση του όρου Ισλαμιστές. Εν πάση περιπτώσει μιλούμε για δύο με τρεις ε, τρομοκράτες οι οποίοι έχουν εκατοντάδες τύπου αγροτικά αυτοκίνητα ε, τύπου το και άλλα, έχουν ε, αυτόματα όπλα, έχουν ε, διάφορα όπλα, διαφόρων διαμετρημάτων, μέχρι και 14-15 χιλιοστών, έχουν RPG, εκτοξευτήρες δηλαδή χειροκίνητους πυράβλων, Με, ένα, με τέτοιες λοιπόν ένοπλες δυνάμεις, σίγουρα εάν δεν ελέγξει κανείς την κατάσταση με πολύ αποφασιστικό τρόπο, σίγουρα αυτό μπορεί να διαρκέσει σε μεγάλο βάθος χρόνου και να ε, οδηγήσει σε μεγάλες καταστροφές. Ο αντίπαλός μας λοιπόν όπως σας είπα είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένος, γνωρίζουν ε, και τους τακτικούς ελιγμούς και πώς να οπισθοχωρούν και πώς να αλλάζουν στόχους στην πορεία και θα έλεγα μάλιστα ε, χρησιμοποιώντας μια στρατιωτική ορολογία, ότι δηλαδή είναι ε, στρατιώτες καλά εκπαιδευμένοι, στρατιωτικοί καλά εκπαιδευμένοι και άρα δύσκολο να ε, περιοριστούν και να τους να τους αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα αναζητούμε πάντοτε το χαμένο χρόνο, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να τον αποκτήσουμε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, ε, προσπαθούμε εν μέρη να επιταχύνουμε όσο το δυνατόν την ε, απλήρη ανάπτυξη και επιχειρησιακή δυνατότητα των αφρικανικών ε, ενόπλων δυνάμεων. Δεχτήκαμε βοήθεια από διαφόρους Ευρωπαίους εταίρους μας και θα ήθελα να αναφέρω τα ονόματά τους γιατί είναι πολύ σημαντικό τα ονόματα των χωρών από πλευράς δηλαδή Βελγίου, Ισπανίας, Γερμανίας, κάτω χωρών, Δανίας, Ηνωμένου Βασιλείου. Ουγγαρίας και Σουηδίας δεχθήκαμε βοήθεια ε, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερο τις χώρες αυτές διότι έθεσαν στη διάθεσή μας μέσα μεταφοράς, στρατηγικά μέσα μεταφοράς για να μπορούσαμε να καλύψουμε αυτή την απόσταση από την Ευρώπη μέχρι την Αφρική και μας ε, ε, έδωσαν και μέσα για να καλύψουμε την απόσταση από το Μαλί στη Σενεγάλη ή από άλλες χώρες προς το Μαλί, Αφρικανικέ, Λάβαμε ιατρικέ ομάδε που θα μα βοηθήσουν. Όλα αυτά μα βοηθούν εξαιρετικά. Εκατοντάδες τόνοι πρέπει να μεταφερθούν και ήδη έχουν μεταφερθεί και αν υπάρχουν και άλλες χώρες που θέλουν εθελοντικά να βοηθήσουν βεβαίως είναι ευπρόσδεκτες. Για να ολοκληρώσω από εδώ θα έλεγα ότι είχαμε ε, και βοήθεια από μη Ευρωπαίους εταίρους, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το παρόν. Επομένως, προσπαθώντα να επιταχύνουμε την ε, ε, σύσταση και την επιχειρησιακή δυνατότητα της αφρικανικής δύναμης ε, και μου θέσατε πολλές ερωτήσεις για, το στρατιωτικό της δυναμικό. Είναι γενικώ ότι η αφρικανική δύναμη δεν έχει ποτέ πολεμήσει μαζί έτσι όπως είναι μια κοινή επιχείρηση ποιο είναι το δυναμικό της, ποιες είναι οι δυνατότητές της. Σίγουρα κάποιες χώρες είναι πιο προηγμένες στρατιωτικά, αφρικανικές, κάποιες άλλες λιγότερο εξαρτάται και από το εκάστοτε πεδίο. Εμείς ως Γάλλοι στρατιωτικοί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι το εξής. Πρώτον, να σταματήσουμε τις επιθέσεις των ομάδων της Τζιχάντ ε, στα κεντρικά ε, σημεία προς τον Μπαμάκο Πρώτον. Δεύτερον, να καταφέρουμε να έρθουν οι αφρικανικές δυνάμεις όσο το γρηγορότερα και να τις εκπαιδεύσουμε, να τις μάθουμε να μπορούν να δρούν και να επιχειρούν στις σωστές συνθήκες, παράλληλα με αυτό που κάνουμε εμείς με τις ένοπλες στρατιωτικές δυνάμεις του Μαλή, το στρατό τον επίσημο του Μαλή, όπου στις πόλεις που κατακτούμε πανακατακτούμε, δίνουμε ε, τη δυνατότητα στο στρατό του Μαλή να ανακτήσει τον έλεγχο των πόλεων αυτό. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο και πολύ χρονοβόρο να σας εξηγήσω όλες τις λεπτομέρειες. Δεν είναι πάντοτε ικανοποιητικά όλα τα ε, αποτελέσματα σε πολιτικό επίπεδο και σε στρατιωτικό, αλλά ε, κάνουμε το παν με τα μέσα που διαθέτουμε. Στις διάφορες ερωτήσεις που μου θέσατε, με ρωτήσατε και το εξής. Πόσο χρόνο θα μπορέσουμε να αντέξουμε μόνοι, εμείς οι Γάλλοι. Πολύ καιρό είναι η απάντηση, παρόλο που δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να είμαστε δύναμη κατοχής. Δεν επιθυμούμε να μην έχει ευθύνες ο στρατός του Μαλή. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βασιστεί κανείς πλήρως σε αυτό το στρατό του Μαλή έτσι στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα. Επομένως, όταν είπα ότι έχουμε την πρόθεση να παραμείνουμε όσο χρειαστεί, αυτό σημαίνει ε, ότι θα παραμείνουμε για όσο χρόνο μέχρι ότου θεωρήσουμε ότι ο στρατός του Μαλή θα είναι πράγματι σε θέση να ελέγξει την επικράτεια, ε, να ε, πάρει τη σκητάλη και να έχει τον έλεγχο των, της επικρατείας του. Τώρα, αν μου ζητήσετε να κάνω μια χρονική εκτίμηση, θα σας δώσω μια χρονική ψαλίδα, αν θέλετε, πολύ ευρεία. Με πάσα ειλικρίνεια δεν, δεν νομίζω ότι είναι λογικό να σας δώσω ημερομηνίες, να σας πω τρεις εβδομάδες, τρεις μήνες ή τρία χρόνια. Θεωρούμε ότι ο στρατός του Μαλή, μάλλον, θα είναι σε θέση να ελέγξει τα εδάφη του ε, μέχρι το τέλος του 2013, μάλλον. Άρα οι αφρικανικές δυνάμεις θα είναι σε θέση να το κάνουν αυτό νωρίτερα. Αυτό εκτιμούμε. Βεβαίως πολλά μένει να γίνουν και αυτές οι αξιολογήσεις θα ενημερώνονται και θα αναθεωρούνται αναλόγως με το πόσο θα προχωρούν οι, οι δυνάμεις οι αφρικανικές και του Μαλή. Άλλο θέμα είναι ότι οι δυνάμει του Μαλή αυτή τη στιγμή πολεμούν τις τρομοκρατικές ομάδες και όσο πολεμούν δεν μπορούμε να τις αποσύρουμε για να τις εκπαιδεύσουμε και να βελτιωθούν. Υπ' αυτή την έννοια πρέπει να ε, ε βρούμε χρόνο και δυνατότητες να στείλουμε άλλες μονάδες που θα πολεμούν για να μπορούμε να εκπαιδεύουμε, για να ξαναμπούν στη μάχη. Τώρα, μήπως θα έπρεπε να στρατολογήσουμε νέους από το μαλλί στρατιωτικούς και στρατιώτες για να τους εκπαιδεύσουμε από το μηδέν. Ίσως και αυτό θα ήταν ε, ε, εξαιρετικά χρήσιμο. Εμείς μπορούμε βεβαίως να ε, κρατηθούμε εκεί για πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό. Στο Αφγανιστάν είμαστε από τα τέλη του 2001, 12 χρόνια. Στη Βοσνία είμαστε από το 92 το πρόβλημα είναι καταρχάς είναι μόνο χρηματοδότηση αν θέλετε. Δεν είναι πρόβλημα αυτό για τις δυνατότητες του γαλλικού στρατού. Τώρα, ως προς τον πληθυσμό ε, του Μαλή, ε, τον τοπικό, ε, φαντάζομαι ότι θα παρακολουθήσατε όλοι τα ρεπορτάζ, τα τηλεοπτικά κανάλια των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη, ο λαός του Μαλή επιθυμεί διακαώς την παρουσία μας εκεί. Είναι πολύ θετική η στάση τους έναντι ημών. Δεν έχουμε πρόβλημα με τον ε, πληθυσμό προς το παρόν. Ως προς τις αλυσίδες χρηματοδότησης των ε, μελών της Τζιχάντ στην περιοχή. Περίπλοκο το ερώτημα, δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να το απαντήσω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ε, το λαθρεμπόριο στην περιοχή ε, είναι ε, πάρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρόν. Μιλούμε για μια περιοχή 6 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιόμετρων, η περίμετρος της Σαχάρα και στην ευρύτερη περιοχή. Σύνορα τα οποία ουσιαστικά είναι αόρατα, είναι νοητά θεωρητικά ε, και δύσκολα τα ελέγχει κανείς. Όπως ξέρετε η φύση μισεί το κενό οι Ιταλοί συνάδελφοι λένε πάντοτε ότι η μαφία ε, εγκαθ και εγκαθίσταται σε ζώνες που δύσκολα ελέγχει το κράτος. Ε, το ίδιο ισχύει και στο Σαχέλ. Είναι μια τεράστια περιοχή ε, ερημική σε πολύ μεγάλο βαθμό, πολύ λίγος πληθυσμός ε, κατοικεί εκεί, επομένως βρίσκουν ευκαιρία εκεί να εδρεωθούν και να επιχειρούν από εκεί. Τώρα, από πού βρίσκουν χρηματοδότηση, αυτό μας ξεπερνά ως στρατιωτικούς, δεν εντάσσεται στο πεδίο της αρμοδιότητάς μας για να είμαι σε θέση να το απαντήσω, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τρόπους να το λύσει το θέμα αυτό. Πώς θα εγγυηθούμε ότι το Μαλί θα γίνει χώρα τρομοκρατών μετά την αναχώρησή μας. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που έχουμε και με το Αφγανιστάν τα τελευταία 12 χρόνια. Θα σας απαντήσω λοιπόν ε, για το τι πιστεύω εγώ ότι θα πρέπει να γίνει. Και μετά βεβαίως οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικοί στις διάφορες χώρες ε, θα πρέπει να αποφασίσουν. Άποψη μου όμως είναι η εξής μετά την αναχώρησή μας. Για να μην γίνει μια χώρα χώρα τρομοκρατών θα πρέπει να υπάρχει νόμιμη κυβέρνηση εξ αρχής εδρεωμένη και ισχυρή δημόσια διοίκηση, δηλαδή να μπορεί η κυβέρνηση να είναι σε θέση να ελέγξει ε, τη χώρα. Και αυτή η πρόταση ουσιαστικά περικλεί ένα ολόκληρο πρόγραμμα μέσα της. Δεν είναι βέβαια υπόθεση στρατιωτικών αυτών, αυτή. Ωστόσο, νομίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διάφορα εργαλεία που μπορούμε να, μπορείτε να αξιοποιήσετε για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δεύτερον, για να μην γίνει μια χώρα χώρα άνδρο ε, τρομοκρατών, θα πρέπει να έχει μια οικονομία, πώς να το πω, ε, νορμάλ. δηλαδή να μην βασίζεται η οικονομία στο ε, λαθρεμπόριο ή να μην είναι ή να μπορεί να είναι αυτάρκη σε κάποιο βαθμό. Και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εργαλεία για να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει η χώρα αυτή για να μην γίνει άνδρο των τρομοκρατών με την αναχώρησή μας να είναι και επίσης αρκετά ασφαλής από την αστυνομική πλευρά ή τη δικαστική ε, πλευρά και βεβαίως και από τη στρατιωτική πλευρά να έχει μια κάποια ασφάλεια έναντι των εξωτερικών απειλών ε, οι οποίες στόχο θα έχουν την ακαιρεότητα των συνόρων της χώρας. Από εκεί και πέρα ε, έχουμε γαλλικές δυνάμεις, έχουμε δυνάμεις του Μαλή και αφρικανικές δυνάμεις, στρατιωτικές. Όλες αυτές οι στρατιωτικές δυνάμεις θα κάνουν το μέγιστο δυνατό ε, με τη στήριξη της Ευρώπης. Υπάρχει όμως και το σκέλος της διακυβέρνησης της χώρας αυτής ε, και το σκέλος της οικονομίας της χώρας αυτής και εκεί οι πολιτικές και όχι οι στρατιωτικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει περισσότερο να επιληφθούν αυτών των δύο θεμάτων. Τώρα, συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. Σίγουρα θα έχετε δει ότι ε, με όλες οι χώρες, οι γύρω χώρες, εκτός από την Αλγερία, γιατί η Αλγερία δεν συμμετέχει στην Αφρικανική δύναμη, όλες αυτές οι χώρες ε, στέλνουν στρατιώτες και στρατιωτικές δυνάμεις στην Αφρικανική στρατιωτική δύναμη, ώστε να συμβάλλουν στην σταθεροποίηση εκ νέου ε, του Μαλή, της χώρας αυτής. Σε γενικές γραμμές δηλαδή, εμείς ως Γάλλοι δεν έχουμε πρόβλημα με την Αφρικανική στρατιωτική δύναμη, η οποία αποτελείται από στρατιώτες από διάφορες αφρικανικές χώρες, τι γύρω αφρικανικές χώρες. Ω προς την Αλγερία, αυτό το οποίο μπορώ να πω και σα το υπενθυμίζω είναι το εξής. Ο ανεφοδιασμός, τα logistics έχουν τεράστια σημασία σε τέτοιου είδου στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι εναέριε μεταφορέ και η Αλγερία έκανε αυτή την τεράστια ε, χειρονομία ε, από πλευράς ε, στρατιωτικής. Μας επέτρεψε, μας άνοιξε τον αναέριό της χώρο. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό δεδομένο, στρατιωτικό δεδομένο. Και αυτό οφείλω να το πω. Συνοψίζοντας λοιπόν, με όλες τις χώρες που βρίσκονται γύρω από το Μαλί και που συμμετέχουν σε αυτή τη διεθνή επιχείρηση, προσπαθούμε να συγκεράσουμε ε, όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουμε για να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή. Ε, προς το παρόν αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η εξέλιξη είναι καλή ως προς την εκοφαντική σιωπή του ΝΑΤΟ, για την οποία με ρωτήσατε. Όπως γνωρίζετε, ε, εκπροσωπώ τη Γαλλία και στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και μπορώ να σας πω ότι δεν τέθηκε επισήμως ερώτημα για το θέμα αυτό από καμία χώρα ε, στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Το συζητούμε στους διαδρόμους, αλλά όχι επίσημο θέμα δεν τέθηκε. Δεν έχει τεθεί. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να ενημερώσουμε τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ για το, τα τεκτενόμενα στο Μαλί. Ο, επι, αρχηγός του Γαλλικού Επιτελείου ε, Ενόπλων Δυνάμεων το έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ καλά πήγαν τα πράγματα. Υπάρχει μια δυσκολία με την Τουρκία η οποία αρνείται ε, την ε, σύγχυση των δύο όρων, δηλαδή την ταύτιση του όρου Ισλαμιστής με τον όρο τρομοκράτης και αν τελικά αποφασιστεί να γίνει πόλεμο στην ε, περιοχή αυτή με το ΝΑΤΟ, τότε σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα με τους Τούρκους. Αυτό το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Τώρα, κατά πόσο υπάρχει δικαίωμα παρέμβασης, ξένης παρέμβασης στο Μαλί, δηλαδή μια χώρα η οποία βρισκόταν ήδη κάπως σε αποσύνθεση, ε, ε, μπορεί κανείς να έχει το δικαίωμα ως ξένος να παρέμβει. Δύσκολη ερώτηση. Εμείς απαγορεύουμε στους εαυτούς μας, εμείς ως στρατιωτικοί απαγορεύουμε στους εαυτούς μας να πάρουμε τέτοιου είδους αποφάσεις. Εσείς έχετε τον μπαλάκι ως πολιτικοί, αν ως πολιτικοί ηθήνοντες εγκρίνετε τέτοιου είδους πράγματα. Για εμάς ως στρατιωτικοί που είμαστε το ερώτημα δεν τίθεται. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε πουθενά χωρίς να έχουμε ε, το πράσινο φως από πλευράς πολιτικών. Και ε, τι ακριβώς συμβαίνει με τις ε, ένοπλες δυνάμεις ΙΠΑ και Καναδά και με την εκπαίδευση εκεί, τις ε, μάχημες αυτές μονάδες. Επέστρεψαν. Ή μάλλον να σας πω, το, διορθώνω, τι συνέβη με τις ομάδες του Μαλή, τις οποίες είχαν εκπαιδεύσει η και ο Καναδάς. Τελικά αποφάσισαν να προσχωρήσουν στους αντάρτες αντί να επιστρέψουν σε εμάς και πώς μπορούμε να ε, ε, εξαλείψουμε πραγματικά την τρομοκρατική απειλή μετά από αυτή την ε, επιχείρηση. Δύσκολο το ερώτημα. Πάλι θα σας πω ότι η φύση απεχθάνεται το κενό. Αν καταφέρουμε να τους διώξουμε πλήρως από το μαλλί, φαντάζομαι ότι θα βρουν χώρο να στεγαστούν σε κάποια άλλη χώρα εκεί γύρω και νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα σε βάθος χρόνου στην ευρύτερη περιοχή και θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί σε βάθος χρόνου. Εκτοπίσεις πληθυσμών. Διαδρομή ανθρωπιστική. Πώς μπορούμε να ασφαλίσουμε τη ΜΚΟ. Νομίζω ότι <clears throat> φυσικά Είμαστε ανθρωπιστές και το έχουμε σκεφτεί. Προσπαθούμε να ασφαλίσουμε τους πρόσφυγες. Θα μεριμνούμε ώστε αυτό να γίνεται πάντοτε στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Δεν είναι καταπληκτικά τα πράγματα, αλλά από όσο γνωρίζω ε, δεν έχουν υπάρξει δεν έχουν υπάρξει ε, αδελφοκτόνες ε, ανάμεσα δηλαδή στους εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες. Στρατηγέ θα χρειαστεί να σας διακόψω γιατί οι διερμηνείς έχουν ε, κάποια ωράρια τα οποία έχουμε ξεπεράσει και θα σας προτείνω να <coughs> συνεχίσουμε στα αγγλικά αν θέλετε. Δεν είστε όλοι γαλλόφωνοι όσοι είστε εδώ, δυστυχώς. Να συνεχίσουμε στα αγγλικά. Εντάξει, δεν το πούμε στο Παρίσι είναι διαταγή αυτή μου δίνετε ή όχι. Μπορούμε να τα πούμε στα γαλλικά, κύριε Πίτσουλα. Μπορείτε να... Ο κύριος Τάνοκ ε, είναι τέλειος γαλλόφωνος, ο, Μίχαελ ε, γαλλικά. Ναι, ο κύριος Τάνοκ μιλάει γαλλικά. Εσείς και εσείς μιλάτε πολύ καλά γαλλικά με την προφορά του Κεμπέκ. Ωραία, συνεχίζουμε στα γαλλικά.